Ladies, gentlemen, Mr. Κυρίες και κύριοι, κυρίες κύριοι και κύριε Κασπάρη και κύριε Καζάκ. Τελείωσε το διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας στο 8, ομάδα εποπτείας, για τον Νότιο Κάφκασο. Υπάρχει μια ομάδα που παρακολουθεί και η οποία συνεδρίασε στις 22 Ιανουαρίου. Πήραν μέρος και οι υπεύθυνοι των τμήματων της Αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης, ο πρέσβης της Αρμενίας και ο πρέσβης της Γεωργίας. Η κυρία Αντρικίενε είναι η η συγγήτριά μας δεν είναι μαζί μας, διότι αν δεν κάνω λάθος έχει πεταχτεί στο Σαντιάγο της Χιλής. Μας άφησε ένα σημείωμα ενημερώνοντάς μας για το τι συνέβη. Ήταν ιδιαίτερος κακοφόρα η συνεδρίαση αυτή η Επιτροπή και οι πρέσβεις επιβεβαίωσαν τη σωστή δυναμική των διαπραγματεύσεων με την Αρμενία και τη Γεωργία τον προηγούμενο χρόνο για τις συμφωνίες FTA. Ο στόχος για την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης μέσα στο 2013 είναι εφικτός και η συγγήτρια είναι ικανοποιημένη γιατί οι δύο αυτές χώρες εξακολουθούν να είναι στραμμένες προς την Ευρώπη. Για το Βιετνάμ τώρα υπάρχει η ομάδα που παρακολουθεί και συνεδρίασε στις 5 Δεκεμβρίου. Πήρε μέρος ο πρέσβης του Βιετνάμ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διευθυντές ε, της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου, η κυρία Κιονίχ. Η συγητής μας είναι η κυρία Ζάχραντιλ λέει ο πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια και αν χρειαστεί θα ε, ακολουθήσει η συζήτηση. Ο κύριος Ζαχραντήλ λοιπόν έχει το λόγο. Να μου επιτρέψετε να σας υπενθυμίσω ότι η συνεδρίαση αυτή συνεδρίασε για πρώτη φορά, συναισθήθη εν πάση περιπτώσει το 2011 Υπήρξε και άλλη μία συμφωνία η οποία συνήφθη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Βιετνάμ, προκαταρκτική. Το 12 υπεγράφηκε αυτή, τον Ιούνιο, στις 22 Ιουνίου του 12. Μέχρι τώρα συνεδρίασε δύο φορές η ομάδα παρακολούθησης και εποπτείας, 5 Δεκεμβρίου η τελευταία φορά, όπως είπατε, ήταν εκεί ο κύριος διαπραγματευτής μας, ήταν ο Βιετναμέζος πρέσβης. Η ενημέρωση για τον πρώτο γύρο των επίσημων διαπραγματεύσεων που έγιναν στο Χανόι ανάμεσα στις 8 και στις 12 Απριλίου, 8 ε, Οκτωβρίου, συγγνώμη, και τώρα ξεκίνησε και ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων από τις 22 ε, Ιανουαρίου μέχρι τις 25. Διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις δηλαδή αυτή τη στιγμή στο, στις Βρυξέλλες. Τίποτα το τρομερό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα. Από ό,τι φαίνεται και από τις δύο πλευρές υπάρχει καλή θέληση Υπάρχει επιθυμία συνέχισης γενικά των επαφών και συζήτησης των προβλημάτων. Είμαστε δεκτικοί και η μεν και η δε και σε σχέση με τα δασμολογικά εμπόδια και πέραν αυτών και στα υπόλοιπα. Μιλήσαμε για το επιχειρηματικό περιβάλλον του Βιετνάμ. Είναι δύσκολο να υπάρξουν βελτιώσεις σε επίπεδο διοικητικό Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα στο μέλλον. Θα δούμε και τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το τέλος της εντολής αυτής. Πάντως μία κάποια πρόοδος προβλέπεται για το 2013 και θα συνεχίσω να σας ενημερώσω. Δεν έχω κάτι άλλο, λέω και ο Σαχράντιλ. Να ευχαριστήσω τους σκιώδεις όλων των πολιτικών ομάδων οι οποίοι ήταν παρόντες στη συνάντηση και οι οποίοι έθεσαν προς συζήτηση πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα με πολύ φιλικό τρόπο, παραγωγικό τρόπο. Πρέπει να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος από το πώς πηγαίνουν τα πράγματα μέχρι τώρα. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Χαίρομαι που βλέπω που οι ομάδες αυτές κάνουν τη δουλειά τους. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια παρατήρηση. Όχι. Οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σημείωσε αυτά τα οποία ακούστηκαν. Δεν υπάρχουν αντιδράσεις από πλευρά της. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο 9. Τριμερής διάλογος. Συνέχιση διαπραγματεύσεων. Ξεκινώντας να πω ότι η εισαγωγική τριμερής διάλογη για το Omnibus 1 διεξήχθη στις 5 Δεκεμβρίου. Μια και η συγγήτρια δεν είναι μαζί μας σήμερα. On this file, uh, that, uh, the next steps are... Τα επόμενα βήματα θα είναι μια εσωτερική συνεδρίαση και μια τεχνική συνεδρίαση που προβλέπεται για τις 26 Απριλίου και επαφή με την εισηγήτρια στις 5 Μαρτίου, μια προκαταρκτική επαφή. Τα πράγματα δεν πάνε γρήγορα. δεν ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να τελειώσουμε έγκαιρα γιατί το πεδίο είναι ευρύτατο. Για τα άλλα δύο θέματα, συγγενικά πνευματικά δικαιώματα και τελωνιακή προστασία, η συγγήτριά μα είναι εδώ και θα της δώσω το λόγο. Η Ζωζέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο που πρέπει να πω είναι ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για την πρόοδο των πραγμάτων. Είναι μια από τις πρώτες εκθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 50, έχουν ξεκινήσει και άλλες τώρα, και είναι η πρώτη φορά επίσης που προσπαθούμε εμείς να ε, διατηρήσουμε τις αποκλειστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής μας, της ΣΥΝΤΑ, σε μια έκθεση η οποία στην αρχή ανήκε στην ΙΝΚΟ, την οικονομική. Υπάρχουν λοιπόν δύο βασικές ιδέες που πρέπει να ελέγξουμε αν θέλετε. Πρόκειται για τα προϊόντα τα οποία μετακινούνται από τη μία χώρα στην άλλη και υπηρεσίες φυσικά και σε επίπεδο διεθνούς συνεργασίας που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής μας Τελωνιακός έλεγχος, δυνατότητες εφαρμογής μέτρων και για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και ταυτόχρονα υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε όλους και το Συμβούλιο και την νομική υπηρεσία και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συνεργασία της, Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Υποθέσεων, μας βοήθησε να ξεπεράσουμε τους δισταγμούς του Συμβουλίου που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στη διεθνή συνεργασία και στην ανταλλαγή ε, μέτρων που είναι απαραίτητο για την καταπολέμηση των πλαστών προϊόντων. Και ο πρόεδρος επίσης ε, της Επιτροπής αυτής ε, έδειξε ότι σέβεται το χώρο της κάθε Επιτροπής. Πολύ ικανοποιητικέ οι εξελίξεις, λέει ο πρόεδρος. Η Επιτροπή πρέπει να κατανοήσει ότι είμαστε φυσικοί σύμμαχοι με αυτήν και έχουμε εδώ ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πώς τα πράγματα εξελίχθηκαν με τον σωστό τρόπο. Ξέχασα να σας πω ότι η ΙΜΚΟ είναι η αρμόδια επί της ουσίας και όχι εμείς. Ένας άλλος τριμερής διάλογος που μας ενδιαφέρει είναι τα εταιρικά μέσα. Και εδώ δεν είμαστε η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή. Η επί της ουσίας επιτροπή είναι η εξωτερικών υποθέσεων εδώ. Η συγγήτρια δική μας είναι η κυρία Ένε, όπως σας είπα είναι στο Σαντιάγο. Και δεν μπορεί να μας πει το τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν ξέρω, ε, θέλετε να γίνει κάποια συζήτηση, έχετε κάποιο σχόλιο, κάποια ερώτηση, δεν φαίνεται. Οπότε για μια ακόμη φορά ευχαριστώ ότι Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκέντρωσε όλα τα στοιχεία τα οποία ήθελε γύρω από το θέμα αυτό, το σημείο 10. Αυτό είναι σοβαρό, βαρύ θέμα θα έλεγα. Πρόσφαση των προϊόντων και υπηρεσιών από τις τρίτες χώρες στην εσωτερική αγορά και στον τομέα των δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων. Πρόκειται για τον κανονισμό της αμοιβαιότητας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Ο κύριος Κάσπαρη έχει το λόγο, δεύτερη ανταλλαγή απόψεων. Έγινε μια συνάντηση ήδη ανάμεσα στον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές και τους αρμόδιους γενικούς διευθυντές της Επιτροπής Εμπορίου και Αγορών και η συζήτηση τώρα θα ασχοληθεί με τις ανησυχίες που εκφράστηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης ανταλλαγής απόψεων. Ο κύριος Κασπάρη έχει το λόγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτός ο φάκελος, τον οποίο σήμερα εξετάζουμε σε δεύτερη ανάγνωση, μας δίνει δύο διαφορετικές θέσεις στην Επιτροπή, οι οποίες ανήκουν και σε διαφορετικές κοινοβουλευτικές ομάδες. Η μία άποψη είναι να απορρίψουμε τελείως τον φάκελο, με την αιτιολογία ότι είναι ένα λάθος σήμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αναφέρεται επίσης ότι και η δική μας αγορά δεν είναι τόσο ανοιχτή όσο θα έπρεπε. Η άλλη άποψη από την άλλη είναι ότι χρειαζόμαστε αυτό το μέσο και νομίζω πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ήδη πάρα πολλούς λόγους για τους οποίους χρειαζόμαστε αυτό το μέσο και η πλειοψηφία έχει αυτή την άποψη. Επιθυμώ να εργαστούμε περισσότερο πάνω στο σχέδιο, σε θέματα ουσίας. Υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε και η πρότασή μου είναι καταρχάς το άρθρο για τις ε, ιδιαίτερα χαμηλές προσφορές. Κατά τη γνώμη μου αυτό το θέμα είναι αρκετά τεχνικό και πιστεύω πως η Επιτροπή ΙΝΚΟ είναι η αρμόδια Επιτροπή για να το επεξεργαστεί και να τους το θεώσουμε, διότι έχουν πολύ περισσότερη εμπειρία από εμά στον τομέα αυτό. Μετά, στα άρθρα 8 και 10, που αναφέρονται επί της ουσίας στο ερώτημα αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από εξέταση μπορεί να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για ε, δημόσιες συμβάσεις σε τρίτες χώρες. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και πιστεύω πως ε, πρέπει να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις ε, λεπτομέρειες, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω πως ε, η αντιμετώπιση όλων μας θα είναι γενικότερα θετική. Το πρόβλημα που έχω είναι στο άρθρο 6 και πιστεύω και πολλοί συναδελφοί έχουν πρόβλημα γι' αυτό. Και η καλύτερη περιγραφή που έχω ακούσει είναι ότι είναι τελείως αυθαίρετο αυτό το άρθρο και πιστεύω πως ε, έχει λίγα πράγματα, έχει λίγη σχέση με την ε, εμπορική πολιτική. Το άρθρο αυτό προβλέπει κάποιες διατάξεις για τις ε, δημόσιες προμήθειες όμως και για τους αναδόχους από τις τρίτες χώρες. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μας έχουν δείξει ότι το άρθρο 6 έχει πρόβλημα. Για παράδειγμα, δύο ή τρία μεγάλα κράτη στην Ευρώπη ε, κάνουν προκήρυξη για νέα βαγόνια για τα τρένα του. Το Βερολίνο, πούμε, για παράδειγμα, στη Γερμανία. Σκέφτεται να χρησιμοποιήσει, για παράδειγμα, το άρθρο αυτό και να δώσει την... Ε, να αναθέσει το έργο αυτό εκτός Υπάρχουν στην περίπτωση αυτή και ορισμένες ε, εταιρείες που έχουν προσφέρει πολύ χαμηλές τιμές, υπερβολικά χαμηλές. Και το ερώτημα είναι στο θέμα αυτό τι θα κάνουμε σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει μέσω του άρθρου αυτού σε ένα κράτος να το χρησιμοποιήσει προς όφελός του, πώς αυτό θα επηρεάσει την εξωτερική πολιτική. Δεν νομίζω πως αυτό θα έχει θετικές συνέπειες. Εάν κάποιο κράτος επιτρέπει στις δημόσιες αρχές του να, κάνουν προσφορές, να δέχονται προσφορές από τρίτα κράτη με υπερβολικά χαμηλές τιμές, πιστεύω πως αυτό λίγο θα προωθήσει την εξωτερική πολιτική. Γενικά, πάντως, το άρθρο 6 είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα. Ένα από αυτά είναι ότι νομικά δεν έχουμε δυνατότητα να ανοίξουμε την ενιαία αγορά για προσφορές από τρίτες χώρες χωρίς πριν να υπάρξει κάποιο σύμφωνο και πιστεύω πως αυτό το επιχείρημα είναι κάτι που θα πρέπει να μας οδηγήσει σε σκέψεις και σε προσπάθειες να το βελτιώσουμε, έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε όλες τις πιθανές εκδοχές. Άλλο ένα πρόβλημα το οποίο έγινε προφανές τις τελευταίες εβδομάδες είναι ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη, τελευταία, έχουν παρατηρηθεί παράνομες ε, συμφωνίες ανάμεσα σε, στο κράτος αυτό και σε τρίτες χώρες και έχει προκύψει η ανάγκη καλύτερης ρύθμισης στις περιπτώσεις αυτές και την δημιουργία μιας δημόσια, ευρωπαϊκής δημόσιας αρχής η οποία θα χρησιμοποιήσει τις καλές πρακτικές και από κοινού θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή εμπορική πολιτική και ρυθμιστικούς κανόνες. Να επαναλάβω, με το άρθρο 6 έχω πρόβλημα, έχω αρκετές αμφιβολίες και όσον αφορά τώρα την διαδικασία. Να σας πω ότι τον Μάρτιο, το Φεβρουάριο μάλλον, έγινε ακρόαση για το θέμα αυτό. Θα γίνει, με συγχωρείτε μάλλον, και ανυπομονώ, μετά οι συντονιστές θα, εξάγουν εκτίμηση επιπτώσεων και σε αυτό το σημείο να καλέσω όλους τους ε, σκιώδεις εισηγητές να συμμετέχουν και να συζητήσουν επί του περιεχομένου. Ελπίζω να το κάνουμε αυτό την ε, επόμενη εβδομάδα, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και να έχουμε αρκετό χρόνο για να προετοιμαστούμε. Μία παρατήρηση ακόμα, κάτι που ακούω πολύ συχνά και δεν είναι δική μας αρμοδιότητα είναι το εξή. τις ε, αμφιβολίες και γενικά τις, ε, ακούω το ερώτημα του πώς αντιμετωπίζουμε εμείς ε, τους επενδυτές από τις τρίτες χώρες, τι γίνεται με αυτούς και με την κατάσταση στην ενιαία αγορά. Αυτή την εποχή βρίσκομαι σε συνομιλίες με αντιπροσώπους εμπορικών συνδέσμων στην Ευρώπη, τους οποίους ανησυχεί η κατάσταση, ανησυχούν για την ανταγωνιστικότητά τους και τη μελλοντική τους ανταγωνιστικότητα και πώς οι προκηρύξεις και η ανάθεσή τους ενδεχομένω σε τρίτες χώρες επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητα στην ενιαία αγορά. Και αυτό επίσης είναι κάτι που θα πρέπει να συζητήσουμε. Το πώς δηλαδή θα προστατεύσουμε την ενιαία αγορά από τον αθέμητο ανταγωνισμό. Τα άρθρα 8 και 10, λοιπόν, συνοψίζοντας με βρίσκουν σε γενικές γραμμές σύμφωνο, διαφωνώ με το άρθρο 6 και κλείνοντας να σας πω ότι ανυπομονώ για τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Ε, το πρωί οι συντονιστές αποφάσισαν να αναθέσουν μία εκτίμηση, να γίνει μία εκτίμηση αυτού του κανονισμού και όσον αφορά την τελευταία σας παρατήρηση, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η ΙΜΚΟ είναι υπεύθυνη και για την εσωτερική πλευρά των δημοσίων συμβάσεων, διότι έχει ζητήσει στην Επιτροπή να αναθεωρήσει τους υπάρχοντες κανονισμούς όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Συνεπώς πρέπει να συντονιστούν οι ενέργειες μεταξύ τους, έτσι συμφωνήθηκε από τους συντονιστές. Τώρα, ο κύριος Σούστεφ, παρακαλώ. Ευχαριστώ τον κύριο Κάσπαρη για τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε το θέμα του. και για τις επαφές που έχει ξεκινήσει με όλους τους της εισηγητές. Κάποια θέματα γενικού χαρακτήρα ακούστηκαν την προηγούμενη φορά και δεν θα χρειαστεί να τα επαναλάβω πάνω στη σημασία που έχει και την ανάγκη που υπάρχει ε, να προωθήσουμε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Γιατί από τη μία θέλουμε να επιβεβαιώσουμε ότι η αγορά μας είναι μια ελεύθερη αγορά αλλά πρέπει να είναι και μια αγορά ε, με ισχύουσα την αρχή της αμοιβαιότητας. Πολλές οικονομίες οι οποίες βρισκόντουσαν στη φάση της ανάπτυξης και έχουν τα πλεονεκτήματα των χωρών που είναι υπό ανάπτυξη δεν έχουν πλήρως αναλάβει τις ευθύνες τους ως μεγάλες οικονομικά ισχυρές χώρες. Αυτά λοιπόν καθιστούν απαραίτητο τον κανονισμό αυτό και σωστή την επιφυλακτικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί. Άρθρο 6 του κανονισμού τώρα θα πρέπει να το εξετάσουμε πιο προσεκτικά. Όπως έλεγε ο Κασπάρη, μπορεί να δημιουργήσει κάποιες ανισότητες σε εσωτερικό επίπεδο. Από την άλλη θα πρέπει και εμείς να σκεφτούμε επί της ουσίας τον τρόπο με τον οποίο θα προστατεύσουμε την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δώσει την δυνατότητα ε, στις αρμόδιες αρχές ε, να εξαιρέσει προτάσεις άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ που το 50% της αξίας των προσφορών αυτών είναι εξωτερικής προέλευσης. Απ' την άλλη θα πρέπει εμείς να μην επιτρέψουμε στις Βεξέλες να λειτουργήσουν ιδιαίτερα συγκεντρωτικά απέναντι στις διάφορες χώρες μέλη. Μιλάμε για κανονισμό, δεν μιλάμε για οδηγία και γι' αυτό αν θελήσουμε να μπούμε σε υψηλό επίπεδο λεπτομέρειας, ε, για το τι θα συμβεί σε κάθε χώρα στην οποία υπάρχουν εντελώς διαφορετικές έτσι και αλλιώς συνθήκες και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο κοινωνικό. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει ουσιαστικό συγχρονισμός. Παρ' όλα αυτά λοιπόν έχουμε προσπαθήσει να πάμε στο βάθος, υπάρχει το πρόβλημα, βλέπουμε ποιες είναι οι δυνατότητες να αποκλείσουμε κάποιες τέτοιες προσφορές, αλλά είναι σαφές ότι καλό θα ήταν να καθαρίσουμε τα κριτήρια μέσω των οποίων σε κάποιες περιπτώσεις θα είναι υποχρεωτικός ο αποκλεισμός αυτός και σε άλλες περιπτώσεις προαιρετικός. Τώρα για το όριο αυτό των άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η Επιτροπή στην πρότασή μας μας λέει ότι μόνο το 7% των προμηθειών έχουν ανώτατο επίπεδο, ανώτερο από τα 5 εκατομμύρια επίπεδο αξίας. Νομίζω ότι αυτό αντιπροσωπεύει το σύνολο της ε, κοινοτικής αγοράς. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι η αξιολόγηση των επιπτώσεων θα μας βοηθήσει να έχουμε περισσότερα στοιχεία σχετικά με την επιλογή του κανοτάτου ή ανωτάτου αν θέλετε αυτού ορίου ανάλογα με τη ροή των ποσών και ανάλογα με την τεχνολογία που προσφέρεται από τις τρίτες χώρες. Ένα τρίτο θέμα είναι οι ιδιαίτερα χαμηλές προσφορές. Εμείς περιμένουμε ακόμα να γίνει η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΙΝΚΟ και μετά στην Ολομέλεια για την οδηγία, για, την κοινή ωφέλεια και τις προμήθειες από πλευράς των οργανισμών κοινή ωφέλειας. Και δεν θα πρέπει το άρθρο 7 να βρίσκεται σε αντίφαση στη συγκεκριμένη περίπτωση με ό,τι ψηφίσουμε στον άλλο κανονισμό. Θα πρέπει να λάβουμε σαφώς υπόψη μας κάποια συγκεκριμένα ανώτατα ή κατώτατα όρια, όπως υποχρέωση ενημέρωσης αναλυτικής, και να υπάρχει και ένα όριο αυτόματο αποκλεισμού για τις υπερβολικά χαμηλές προσφορές. Η Επιτροπή ΙΝΤΑ έχει εκφραστεί επ' αυτόν όταν εμείς ε, εκδώσαμε τη δική μας ε, γνωμοδότηση σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες ε, και ιδιαίτερα για τον τομέα της κοινή ωφέλεια. Τώρα για τα εισαγόμενα από τις τρίτες χώρες. Δεν πρέπει να εφαρμόζουμε τα ίδια μέτρα με τις φτωχές χώρες, με τις υποανάπτυξη χώρες, χώρες με οικονομίες που δεν είναι μόνο αναδυόμενες αλλά έχουν πλέον πλήρως αναδυθεί. Ένα τελευταίο σημείο αφορά τις έρευνες και τις διαβουλεύσεις. Σχετικά με το κεντρικό σημείο, θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία ενός μηχανισμού έρευνας και διαδοχικών διαβουλεύσεων, ξεκινώντας από τις διαδικασίες αντι-dumping εις βάρος τρίτων χωρών. Η φάση αυτή θα κλείνει με την επιβολή περιοριστικών μέτρων στα πλαίσια της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά. Θεωρώ παρόλα αυτά ότι η διάρκεια των ερευνών θα πρέπει να μειωθεί και θα πρέπει να διευκρινιστεί καλύτερα η λογική διαδοχή, αν θέλετε, των ακολουθούμενων φάσεων, έτσι ώστε να αφήσουμε καθυστερήσεις από πλευράς τρίτων χωρών που έχουν εμπλακεί σε διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Μήπως μπορώ όσον αφορά την ε, μελέτη επιπτώσεων να επανέλθω στο σιώδη Ζητώ συγγνώμη. Η Επιτροπή πρώτα. Είναι έτοιμη η Επιτροπή. Είμαστε στη διάθεσή σα, κύριε Πρόεδρε. Αν θέλετε, μπορούμε να μιλήσουμε τώρα ή αργότερα. Ό,τι προτιμάτε. Πρώτα να ακούσετε τι ερωτήσει, ό,τι θέλετε. Πρώτα θα ακούσουμε του σκιώδει και μετά εσεί. Ευχαριστώ πολύ. Κατόπιν, με την Καζάκα, παρακαλώ, σκιώδη συγητή. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες εδώ. Νομίζω ότι πολλά που έχουν σχέση με την αποτελεσματικότητα του σχεδίου κανονισμού έχουν ήδη αναφερθεί από τον εισηγητή και ήδη συζητήθηκαν όταν έγινε η πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Αλλά πιστεύω ωστόσο ότι υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Συμφωνώ με τον στόχο αυτού του σχεδίου κανονισμού, αλλά όχι με τη διαδικασία που προτείνεται. Ο κύριος στόχος αυτού του σχεδίου κανονισμού, όπως γνωρίζουμε, είναι να επιστήσουμε την προσοχή των ατόμων στις ε, τρίτες χώρες, παροτρύνοντάς τους να υιοθετήσουν τους ίδιους κανόνες ε, για τις κρατικές προμήθειες, τις Δημόσιας συμβάσεις. Αλλά υπάρχει η τάση ότι αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως προστατευτισμός. Τώρα, κατά πώς θα λειτουργήσει αυτός ο κανονισμός, θα το δούμε αν θα οδηγήσει σε ένα άνοιγμα ε, των αγορών των τρίτων χωρών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με απασχολεί το θέμα ότι μπορεί τελικά να έχουμε την τάση να κλείσουμε την αγορά. Πρέπει να βρούμε τους μηχανισμούς που θα επιτρέψουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές αυτές. Τα άρθρα 9 και 10 αφορούν αυτό το αντικείμενο. Και πιστεύω ότι πρέπει να ασκήσουμε πίεση σε αυτές τις χώρες που δεν ανοίγουν τις αγορές τους σε μάς Και πρέπει να παρατηρούμε αυτές τις χώρες να θεσπίσουν μέτρα βιότητας. Αλλά αυτή η προσέγγιση οδηγεί την Επιτροπή ε, σε μια συνεργασία με τις τρίτες χώρες, σε μια προσπάθεια εναρμόνισης ε, των εμπορικών μας πολιτικών. Η Διερμηνέα λέει ότι δεν ακούει ε, τον ομιλητή επειδή δεν ακούει το μικρόφωνο του. Επειδή το μικρόφωνο του Προέδρου συγχρόνως. αλλά τελικά μπορεί αυτά τα οποία κάνουμε να έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Εάν αποκλειστούν ορισμένοι προσφέροντες, και αυτό επαφείεται στη διακριτική τους ευχέρεια, αλλά όλα αυτά δεν νομίζω ότι οδηγούν στη θέσπιση κοινών κανόνων Ας πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα. Ας πούμε ότι υπάρχει μια προκήρυξη για δημόσια σύμβαση στο Λονδίνο και μια άλλη στην Πρατισλάβα και υπάρχει μια κινέζικη εταιρεία που προσφέρει στη μία περίπτωση και μια άλλη κινέζικη εταιρεία προσφέρει στην άλλη περίπτωση. Η μία αποκλείεται και η άλλη όχι. Δεν είναι σαφές γιατί μία εταιρεία γίνεται αποδεκτή και όχι άλλη. Θα ήταν προτιμότερο να ανοίξει η αγορά των δημοσίων συμβάσεων, θα ήταν προτιμότερο να ανοίξει η αγορά των δημοσίων συμβάσεων ε, στη μία χώρα και όχι στην άλλη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Διότι δεν θα πρέπει να έχουμε διαφορετικούς κανόνες, άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Η διαδικασία του άρθρου 6 πρέπει να αναθεωρηθεί για να υπάρξει πραγματική εναρμόνιση που θα επιτρέπει την πραγματοποίηση των στόχων αυτού του σχεδίου κανονισμού. Ευχαριστώ. Next, The Greens. Κύριε από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Πράγματι, αυτό το θέμα δεν είναι εύκολο διότι δημιουργεί αντιδράσεις και μέσα στο Συμβούλιο και αμφιλεγόμενες θέσεις στα πλαίσια του Κοινοβουλίου. Το πρώτο θέμα επί του οποίου υπάρχει διαφωνία είναι ότι σήμερα δεν έχουμε όλα τα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να κρίνουμε κατά πόσον αυτό το προτινόμενο μέσο είναι το σωστό, το κατάλληλο. Και η μελέτη επιπτώσεων που προτείνει η Επιτροπή μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, πιο λεπτομερείς πληροφορίες, για παράδειγμα, σχετικά με το ποσοστό δίσδυσης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε εξωτερικές αγορές και το αντίστροφο. Ε, τη θέση που έχουν οι εξωτερικές επιχειρήσεις ε, χωρών, όχι μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις δικές μας αγορές. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο σημείο το οποίο μου φαίνεται πιο σημαντικό, πιο ουσιαστικό θα έλεγα. Το λέμε καθημερινά, το έχουμε ήδη πει, καθημερινά το διαβάζουμε σε εφημερίδε. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πολύ του συμπολίτε μα. Αντιμετωπίζουμε μια πολύ σημαντική οικονομική κρίση με μια διαδικασία αποβιομηχανοποίηση που ανησυχεί του πάντε. Και τη στιγμή που μιλάμε για 18% του ΑΕΠ της Ευρώπης, όπου μιλάμε για δημόσιο χρήμα, σε αυτή την πρόταση μιλάμε μόνο για εμπόριο. Φυσικά βλέπουμε τη Βούλη της Επιτροπής να αποκλείσει κάθε πιθανότητα χρήσης των δημοσίων συμβάσεων από εθνικές ή τοπικές αρχές για σκοπούς βιομηχανικής πολιτικής ή επίτευξης δημοσίων σκοπών στόχων που είναι απόλυτα θεμητή και βλέπουμε τη βούληση της Επιτροπής να περιορίσει τις δυνατότητες παρέμβασης για υπηρεσίες και αγαθά που δεν καλύπτονται. Αλλά αυτή είναι μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση, δηλαδή να δούμε κατά πόσο το διακύβευμα στις δημόσιες αγορές αφορά μόνο αφενός τα όσα υπάρχουν στην εσωτερική αγορά, δηλαδή η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα των δαπανών, αν θέλετε, υπό την έννοια του να βρει κανείς το μειοδότη. Και όταν μιλάμε για διεθνέ εμπόριο, να έχουμε ω μόνο κριτήριο, μοναδικό κριτήριο, την αμοιβαιότητα. Για παράδειγμα, βλέπουμε όταν δούμε τι γίνεται με ε, την οδηγία για τη, ε, του οργανισμού κοινή ωφελία, βλέπουμε θέματα κοινωνικά. Στα άρθρα 58 και 59 υπάρχουν τα κοινωνικά διακυβεύματα που έχουν σχέση με τις εμπλεκόμενες χώρες. Ε, ε, αλλά εδώ πέρα δεν θέλουμε να μιλάμε για κοινωνικά διακυβεύματα, για στόχους δημοσίας ε, πολιτικής ή τοπικής πολιτικής. Δεν υπάρχει θέμα να παρεμβαίνουμε σε θέματα της βιομηχανίας στην Ευρώπη. Τι θέλουμε τη βιομηχανία στην Ευρώπη και ε, τι προβλέπουμε μετά από 10, 5, 10, 15 χρόνια και σε τι οι δημόσιε συμβάσει μπορούν να είναι χρήσιμε. Απλά και μόνο περιοριζόμαστε στο θέμα τη αμοιβαιότητα. Και αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ οριακό. Είναι θεμητό μεν, αλλά είναι οριακό. Θα ήθελα κάποια στιγμή, ειλικρινά, να γίνει αυτή η συζήτηση η μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση, δηλαδή σε τι μα χρησιμεύουν οι ε, κρατικές προμήθειες και δημόσιες συμβάσεις. Ε, φυσικά πρέπει να υπάρχει διαφάνεια ε, πρέπει να είναι αποτελεσματικέ όσον αφορά τι δημόσιε δαπάνε. Αυτό είναι απόλυτα προφανέ και πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα μεταξύ κοινωνικών εταίρων. Αυτό πάλι είναι προφανέ. Αλλά όταν μιλάμε για δημόσιο χρήμα που αφορά το 18% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ σε μια μεγάλη οικονομική κρίση, το να σταματήσουμε εκεί, αυτό πιστεύω ότι είναι πραγματικά οριακό. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της ομάδας ECR. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω πως η σύνοψη του Ντάνιελ ήταν εξαιρετική. Τι θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει δουλειά. Όλοι αυτό θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ντάνιελ, ανέφερε κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Μίλησε για την εσωτερική αγορά εκτός από την εξωτερική αγορά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το Ηνωμένο Βασίλειο πρόσφατα ε, δημιούργησε μια προσώστοση για τις μεγάλες ε, δημόσιες προμήθειες και μια χώρα ανέλαβε το social engineering, όπως το λέμε, και σε περίπτωση, και, δηλαδή, αυτό τι σημαίνει, ότι σε περίπτωση που γίνει δεκτή η προσφορά, πολλοί κόσμος θα μείνει άνεργος. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι τι γίνεται με τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα όρια όχι μόνο στην εσωτερική αγορά, αλλά και με τον ανταγωνισμό εκτός αγοράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαιρετική είναι η έκθεση και είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσουμε σε πολλά σημεία με τον Ντάνιελ διότι το θέμα είναι σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Χέλμουτ από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ συμφωνώ με τους προλελήσαντες. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Παίζονται πολλά. Πρέπει να δούμε πώς θα ασχοληθούμε με τις επιμέρους λεπτομέρειες και πώς θα τις ε, συνδέσουμε. Είτε θα πούμε ότι συμφωνεί κατά βάση με την προσέγγιση μας, αλλά θέλουμε να δούμε τις λεπτομέρειες, είτε διαφωνούμε και πρέπει να προτείνουμε λύση. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις, ιδιαίτερα με το άρθρο 8, ανάμεσα στον εισηγητή και στην δική μας ομάδα. Με το άρθρο 6 όμως έχουμε παρόμοιες απόψεις με τον εισηγητή και θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Τι θα γίνει με τις ε, δημόσιες ε, προκήρυξεις, τι θα γίνει με τις ε, παραχωρήσεις. Αυτά τα ερωτήματα με οδηγούν στο να πω ότι καλό θα ήταν να δώσουμε και στην Επιτροπή των Περιφερειών το φάκελο αυτό για να γνωμοδοτήσει και επίσης να ληφθούν υπόψη και άλλα αντικειμενικά κριτήρια, καθώς και ο κίνδυνος της εμπορική δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αποκλειστεί ο κίνδυνος μέσω επιδοτήσεων και να υπάρχει έλεγχος στις διαδικασίες των προκηρύξεων. Μετά, Πώς θα αντιμετωπίσουμε το άνοιγμα της αγοράς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, παγκόσμια. Πώς θα εισχωρήσουμε στις αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά, τα συνδικάτα έχουν έντονες ανησυχίες, διότι διακυβεύονται θέσεις εργασίας και το συζητήσαμε. Το ερώτημα είναι πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα του dumping, του κοινωνικού dumping και των dumping των μισθών, των απολαβών. Την χειροτέρευση των συνθήκων εργασίας εν μέσω της οικονομικής κρίσης. Αυτό πρέπει να υπάρχει στην έκθεση. Το Γερμανικό Συνδικάτο Βέρντι έχει καταστήσει σαφές ότι ακόμα ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, μια, για έναν έλεγχο, για μια ελεγκτική αρχή, θα είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση, θα αποτελέσει υπόδειγμα αυτή η αρχή ελεκτική. διότι το θέμα δεν είναι η καλύτερη προσφορά, η χαμηλότερη προσφορά. Δεν θέλουμε η καλή συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού φορέα να είναι η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας. Δεν θα μακρηγορήσω περισσότερο. Μία παρατήρηση να κάνω κλείνοντας πρέπει να ασχοληθούμε με το θέμα των αγαθών και των υπηρεσιών και των δασμών και να φροντίσουμε να ασχοληθούμε με το ζήτημα της διαφάνειας. Εμείς θα εργαστούμε εντατικά για την έκθεση αυτή και θα συνεισφέρουμε όσο μπορούμε για να βελτιώσουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο, πιστεύω. Μάλιστα. Δεύτερος γύρος. Κυρία Νάρα Μπέρ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σιγητή, χαίρομαι πολύ για αυτή την πρωτοβουλία που ανέλαβε ο κύριος Μπανί, που σταθμίζει ορισμένα ουσιαστικά θέματα όσον αφορά την ισορροπία των διεθνών ανταλλαγών και την ενότητα που μπορεί και επιθυμεί να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ των εταίρων της. Σχετικά με τις διαβουλεύσεις που οργανώθηκαν, βλέπουμε ότι ήδη οι οικονομικοί παράγοντες είναι υπέρ μιας δράσης της Ένωσης μέσω ενός νομοθετικού μηχανισμού. Παρόλο ότι αυτό πολλές φορές ελέγχθη, δεν πρόκειται για μέτρα προστατευτισμού από τη δική μας άποψη τουλάχιστον, αλλά πρόκειται εδώ ε, για την προσπάθεια να ανταποκριθούμε στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν το 50% των δημοσίων συμβάσεων στον κόσμο, επειδή είναι κλειστέ αυτέ οι δημόσιε συμβάσει στι ευρωπαϊκέ αγορέ λόγω προστατευτισμού ή δεσμολογικών προτιμήσεων, ε, λαμβάνοντα υπόψη ε, το πλαίσιο. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειε, απλά και μόνο ορισμένε παρατηρήσει όσον αφορά το πραγματικό πρόβλημα το οποίο θέλουμε να λύσουμε η υπόθεση από οποία βασίζεται αυτό το μέσο είναι ότι οι δημόσιε συμβάσει τη Ευρώπη είναι πιο ανοιχτέ στι ξένε επιχειρήσει από ότι το αντίστροφο. Οι ξένε δηλαδή επιχειρήσει ανοιχτέ στι ευρωπαϊκέ. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε 80% ε, ανοίγματο στα πλαίσια διεθνού Συμφωνίας, έναντι 12% στι ΗΠΑ ή 4% τη Ινδίας. Αλλά πιθανόν χρειάζονται περισσότερα στοιχεία ε, να στηρίξουν αυτές τις σκέψεις μας και γι' αυτό θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποιο είναι το ποσοστό των δημοσίων συμβάσεων που έχουν αναλάβει ε, έχει ανάβει η Ευρώπη από ε, επιχειρήσει με τις τρίτων χωρών με τις οποίες δεν έχουμε σύμβαση και το αντίστοιχο πόσες δημόσιες συμβάσεις έχουν παράσχει αυτέ οι ξένες επιχειρήσεις τις ευρωπαϊκές. Δεύτερο, η λύση η οποία έχει προτιμηθεί. Έχει προτιμηθεί εδώ η θέσπιση ενός νομοθετικού μηχανισμού και όχι το soft close. Δεν αποκλείσατε ε, το Buy the Plan Act για τις ε, αγορές που καλύπτονται όπως ε, στην Ινδία και στις ΗΠΑ, αλλά αυτό μπορεί ε, να δημιουργήσει προβλήματα στους μηχανισμούς που θέλετε εσείς να καταργήσετε. Χωρίς να προδικάσω το τι θα συμβεί, πιστεύω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις που θα έχει αυτός ο μηχανισμός, αυτοί οι μηχανισμοί μάλλον, και να δούμε τι έχετε να μας πείτε πάνω σε αυτά τα θέματα κατόπιν για ε, τους κανονισμούς καταγωγής που ισχύουν Πώς μπορεί ένα θέτος αρχή να πιστοποιήσει την καταγωγή ε, των μέσων, αν προέρχονται από τρίτες χώρες, ε, κατά 50% των τμήματων που απαρτίζουν αυτό το μηχάνημα, τη στιγμή που δεν ξέρουμε ε, από πού προέρχονται αυτά τα μηχανήματα. Ένα άλλο σημείο το οποίο αφορά τις έρευνες. Νομίζω ότι πρέπει να φροντίσουμε αυτέ οι έρευνε που προβλέπονται στο άρθρο 6 και 9 του κανονισμού να μην διαρκούν για πάντα. Κυρίως όταν το επίπεδο πρόσβασης ε, ε, στην αγορά μιας τέτοια χώρας είναι γνωστό από προηγούμενη έρευνα. Εδώ δεν θα πρέπει ε, να δούμε γιατί να θεωρούμε ότι η, απάντηση η μία απάντηση από την Επιτροπή είναι ρητή αποδοχή. Τώρα, όσον αφορά το, όσο προβλέπονται στο άρθρο 10, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι η βάση αυτού του άρθρου και όσον αφορά τις χώρες με τις οποίες ε, υπάρχουν διαπραγματεύσεις, δεν θα πρέπει να καθορίσουμε ένα όριο, ένα χρονικό όριο όταν οι διαπραγματεύσεις ε, δεν προχωράνε. Αναφέρομαι εδώ κυρίως στην Ινδία ή τη Ιαπωνία. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ. Τέλος. Έμα Μαρκάκη, σκιώδης ζητώ συγγνώμη που δεν σα έδωσα το λόγο πρωτήτερα. Ε, Ξεφνικά κατάλαβα ότι είχα ένα μανδύα που με έκανε αόρατη σήμερα το απόγευμα. Από εδώ και πέρα με βλέπετε πρόεδρε οι συζητήσεις που έγιναν ανάμεσα στις πολιτικές ομάδες ήταν θετικές. Και ήταν εξαιρετικός ο κύριος Κασπάρη σε επίπεδο συντονιστικό. Υπάρχουν όμως και αρκετές διαφορές πάνω στην πρόταση αυτή. Σε βασικά θέματα. Υπάρχει μια πλειοψηφία υπέρ των προτάσεων και μιας περισσότερο ιδεολογικής στάση. Αν θα πρέπει να εξετάσουμε δηλαδή αν το μέσο αυτό είναι το κατάλληλο μέσο ή αν δημιουργεί κάποια από τα προβλήματα τα οποία υποτίθεται καλύτερα να αντιμετωπίσει. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί λοιπόν πριν νομοθετήσουμε και γι' αυτό οι συστάσεις του εισηγητή να προχωρήσουμε σε μια λεπτομερή αξιολόγηση των προτάσεων από το Κοινοβούλιο είναι κάτι το απαραίτητο. Εμείς πιστεύουμε στο κοινοβούλιο μας ότι παρόλο τον έλεγχο που έχει γίνει σε επίπεδο με τη μελέτη επιπτώσεων της Επιτροπής, πρέπει να είμαστε απόλυτα ενημερωμένοι σχετικά με τις συνέπειες πριν προχωρήσουμε σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Είχαμε στις 8 Ιανουαρίου μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώς οι συνάδελφοι δεν ήταν παρόντες, ο κ. Κάσπαρη όμως και εγώ ήμασταν εκεί. Και ήταν αποκαλυπτικές οι συζητήσεις που είχαμε είχε ζητήσει από τον Μάρτιο του 12 τη γνωμοδότηση της νομικής τους υπηρεσίας, αλλά επειδή είχαν κλείσει για διακοπές μετά και επειδή είχαν πάρα πολλές ανησυχίες γενικότερα, είχαν μεν ε, εφησυχάσει σε σχέση με τη διόρθωση των ανησυχιών αυτών, και παρόλες τις ε, γνώμες της νομικής υπηρεσίας ε, μειώθηκε το ανώτατο ή κατώτατο όριο αν θέλετε από τα 10 εκατομμύρια στα 5 εκατομμύρια. Ανησυχώ πάντως για την πρόταση αυτή. Θεωρώ ότι η πρόταση αυτή θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορώ σε αυτή τη φάση να υποστηρίξω το προτινόμενο μέσο μείωσης γενικά στις αγορές μας ε, από πλευράς προϊόντων και υπηρεσιών από τρίτες χώρες. Αυτό είναι αρνητικό. Και ακόμα και αν δεν επηρεάσει αρνητικά και δεν οδηγήσει στο κλείσιμο της κοινοτική αγοράς, το προτινόμενο μέτρο είναι σαφές ότι μπορεί να οδηγήσει έμεσα στο κλείσιμο των εθνικών αγορών. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε πού βρισκόμαστε τώρα, σε ποια φάση είμαστε, γιατί υπάρχει κίνδυνος ιδιαίτερα το άρθρο 6 να χρησιμοποιηθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να παραταθεί η κατάσταση προστατευτισμού που ισχύει. Και αυτό είναι αντίθετο με την υποχρέωσή μας για να ανοίξουμε τις αγορές στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου. Δεν ξέρω αν σε αυτή τη φάση μπορούμε να θεωρήσουμε χρήσιμη μια συζήτηση η οποία αναφέρεται στο μακρινό μέλλον. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να ακολουθήσουμε το δρόμο αυτό ο οποίος προτείνεται. Παίζουμε με τη ζωή των ανθρώπων, παίζουμε δηλαδή με τις εργασίες, τις θέσεις εργασίας των ανθρώπων και θα πρέπει να συνεχίσουμε με πάρα πολύ επιφυλακτικότητα και να σταθμίσουμε επίσης πολύ επιφυλακτικά τις ε, δυνατότητες που ανοίγονται μπροστά μας. Έχουμε ένα πρόβλημα, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, πρέπει να ψηφίσουμε τώρα. είναι ιερός όπως ξέρετε ο χρόνο της ψηφοφορίας και δεν έχουμε κλείσει ακόμα τη συζήτηση αυτή. Πρέπει να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την αντίδραση επίσης και του εισηγητή. Και γι' αυτό παρακαλώ ζητώ να διακόψουμε, να ψηφίσουμε και να επανέλθουμε αμέσως μετά. Καλώς λοιπόν. Ας περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία. Αυτόν που έχουμε να ψηφίσουμε, το πρώτο, είναι το 12. Are you ready? Okay. Item 11. 12, 12. 12, sorry. Το 12 λοιπόν. I, δικαίω μπορώ να προσθέσω τις ψήφους αυτών που ξέχασαν την κάρτα τους, εφόσον μου το πούνε βέβαια. το πρώτο θέμα είναι η θέση μας σχετικά με την δεύτερη ανάγνωση του κανονισμού για πρόσβαση στην αγορά. Πρέπει να διαβάσω την απόφαση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν σε ανεπίσημες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή για να φτάσουμε σε μια συμφωνία για τη δεύτερη ανάγνωση το νομοθετικό ψήφισμα της 13 η Σεπτεμβρίου του 2012 θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για την εντολή της διαπραγματευτικής ομάδας. Και η διαπραγματευτική ομάδα θα αποτελείται από τον πρόεδρο, τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές. Ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν. Α, η, ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν. Ψηφίζεται. πέρα της ψηφοφορίας. 23 υπέρ. 24 υπέρ, 2 κατά μία αποχή. Περνάμε τώρα στο άρθρο υπαρίθμου 13. Ψηφοφορία της νομοδότησής μας προς την Επιτροπή ΔΕΒΕ για την πρόθεση της ανάπτυξης μέσω του εμπορίου. Δύο ξεχωριστές εκθέσεις, μία από εμά μία από αυτούς και κάθε μία θα γνωμοδοτήσει και για την έκθεση της άλλης επιτροπής. Ψηφίζουμε λοιπόν όχι τις, την έκθεσή μας αλλά την γνωμοδότησή μας για την έκθεση τους. Υπάρχουν 42 τροπολογίες. Θα ξεκινήσω με την τροπολογία υπαριθμένα. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 1 υπέρ, δεκτή. Τροπολογία 6, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2. Ποιοι είναι υπέρ. Δεκτή. Η 11. Έκανα λάθος λέει ο πρόεδρος. Η 12 λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Δεκτή. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 25 ψηφίζεται. Τέλος. Απερίφθη. 26 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 27 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 28 υπέρ, συγγνώμη, 28 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 29 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Όχι, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 29. Τέλος. Απερίφθη. 30. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 31. Υπέρ, κατά, αποχές. Το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Θα λάβω υπόψη μου και τη δική σας ψήφο. Τέλος της ψηφοφορίας. Υπάρχουν δύο επιπλέον ψήφοι, συνεπώς περνάει η τροπολογία. Δεκατέσσερις κατά, δεκαπέντε υπέρ εννοεί ο πρόεδρος. Τροπολογία 32 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 36 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 37. Σε δύο τμήματα η 37. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 38 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Καλώς, τότε ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 38. Τέλος της ψηφοφορίας. Σκίνερ και Ζαντό, ναι ή όχι. Ναι, το ίδιο αποτέλεσμα, 15 υπέρ, 14 κατά. Συμβιβαστική 6 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, ποχές δεκτή. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, ποχές δεκτό. Συμβιβαστική, ή μάλλον τροπολογία 42 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Τελική ψήφος τώρα. Ηλεκτρονική ψήφος, τελική, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. 20 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Υπολογίζουμε και την ψήφο του κύριου Σκίνερ. 8 αποχές. Επόμενο θέμα. 14. Κριστιανά Μουσκαρδίνη, συγγήτρια για την βιωσιμότητα στο πλαίσιο της παγκόσμιας αλυσίδας αξίας του βαμβακιού. Σύνολο υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16, υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Να κοιτάξουμε τη 16 ηλεκτρονικά. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 15 ψήφοι υπέρ, 12 κατά, μία αποχή, εγκρίνεται. Επόμενη τροπολογία 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 21. Άρχεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 21. Πέρας ψηφοφορίας. Όλοι ψήφισαν με τις κάρτες. Εγκρίνεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24. Υπέρ. Κατά να κοιτάξουμε την 22 ηλεκτρονικά, ωραία. Ας ψηφίσουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 24. 24, τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Εγκρίνεται. Νόμιζα ότι το ΕΛΚ ψηφίζει, καταψηφίζει πάντα την κυρία Κέλλερ. Τροπολογία 27 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 30, εγκρίνεται. 33, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τη 31. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 34. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, Αποχής απορρίπτεται. 38 υπέρ, κατά, Αποχής απορρίπτεται. 39. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 40 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Αιτιολογικές σκέψεις. Τροπολογία 6. Πολ Υπάρχουν αντιρρήσει στην ψηφοφορία των προφορικών τροπολογιών. Δεν απορρίπτονται. Α ψηφίσουμε λοιπόν. Τροπολογία 6. Προφορική υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για την 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 8. Προφορική τροπολογία. Ας ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 13. Χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Citations τώρα. Το πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οριστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 30. Με 27 ψήφους υπέρ, μία αποχή, καμία ψήφο υπέρ. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ας καθίσουμε. Ήσυχα παρακαλώ και γρήγορα. Let's Ας καθίσουμε λοιπόν. Σας παρακαλώ, καθίστε. Παρακαλώ, ησυχία, το λόγο θα δώσουμε στην Επιτροπή σε λίγο. Λίγο σεβασμό. Λίγο σεβασμό να επιδείξετε και για την Επιτροπή και για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που περιμένατε το σύνορα. Έχετε το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά για μας να πούμε δύο λόγια. Δηλαδή να παρουσιάσουμε την ε, εκτίμηση επιπτώσεων και να τη συνδέσουμε με τα όσα ακούσαμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας πω, και αυτό δεν είναι μυστικό, ότι αυτή η αξιολόγηση επιπτώσεων αντικτύπου υπήρξε πολύ δύσκολη για μας ήταν η βάση απόφασης της Επιτροπής. Γι' αυτό τελικά όλοι ήταν πολύ ικανοποιημένοι, συμπεριλαμβανομένοι και της νομική υπηρεσία. Αυτά είναι τα εσωτερικά μας θέματα. Η συζήτηση κατέδειξε ήδη ότι τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αντιμετωπίζουμε στην μελέτη αντικτύπου και στις άλλες μελέτες αντικτύπου πρέπει να δούμε είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να δούμε και αν υπάρχει τεχνική συζήτηση που επιθυμείτε να γίνει για να επισέλθει σε λεπτομέρειες, μπορεί να συμβεί. Καταρχήν ο ορισμός του προβλήματος είναι φανερό ότι αν θέλετε να εκτιμήσετε ποσοτικά αυτά τα θέματα, μπορεί να γίνει για προβλήματα, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση αυτό ήταν σχεδόν αδύνατον. Επειδή δεν υπάρχει συστηματική υποβολή αναφορών για τις ξένες προσφορές. Υπάρχουν ε, ορισμένες προσφορές που γίνονται εντός Ευρώπης, δεν θεωρούνται ως ξένες αλλοδαπές. Λοιπόν, ε, όταν οι επιχειρήσεις της Ευρώπης κάνουν προσφορές στο εξωτερικό, δεν μας το αναφέρουν. Λοιπόν, δεν έχουμε, δεν έχουμε στοιχεία για το πότε κάνουν προσφορές και αν έχουν απορριφθεί αυτές τις προσφορές. Συνεπώς θα δείτε στη δική μας τη μελέτη υπάρχουν στοιχεία που έχουν σχέση ε, με ε, τις συμβάσεις που ξεκίνησαν το 2005 και ορισμένες εκτιμήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται, εκτιμήσεις που δείχνουν ένα πράγμα τουλάχιστον. Ότι ε, υπάρχει άνοιγμα αγορών που μπορεί να εκτιμηθεί ποσοτικά. Εμείς προσφέρουμε ε, ένα δισεκατομμύριο περίπου σε ποσά προσφορές που μπορούμε να ανοίξουμε σε άλλες χώρες. Λοιπόν, θα πρέπει να μας πούν πόσες προσφορές έχουν γίνει και να δούμε κατά πόσον υπάρχει ποσοτική εκτίμηση που μπορεί ε, να υπάρχει και αν έχετε το δικαίωμα να κάνετε προσφορές για ορισμένες δημόσιες συμβάσεις. Ε, περίπου έχουμε 50 δισεκατομμύρια εμείς, ε, οι Αμερικανοί είναι λιγότερα και για Ιαπωνία ας πούμε 27 δισεκατομμύρια και ούτω καθεξής, θα τα δείτε. Τελικά όμως δεν θέλουμε να κρίνουμε σε άλλες χώρες, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να σας πούμε πόσες δεσμεύσεις υπάρχουν. Αυτό μας λέει η μελέτη αντικτύπου ανά κλάδο και κατόπιν λέει που είμαστε δυνατοί Ακούσαμε ότι ε, υπάρχει ένας κύκλος εργασιών 3-5%. Αυτό αντίκειται προς την πρότασή μας. Όχι, είναι ένα επιχείρημα το οποίο εξηγεί ότι υπάρχουν πολλοί περιορισμοί και νομικοί περιορισμοί. Τι μπορούμε να κάνουμε από πολιτική άποψη, να βρισκόμαστε, σε, να βρισκόμαστε ίσοι όρες με τους άλλους. Θέλουμε λοιπόν αυτή η ποσοτικοποίηση, αυτή η μελέτη αντικτύπου να μας φέρει σε ένα ισότιμο επίπεδο. Δεν μπορούμε ποτέ να πούμε ότι αν γίνει αυτό, τότε ε, θα μας ανατεθούν περισσότερες συμβάσεις ή θα κερδίσουμε περισσότερα χρήματα έχουμε, μπορεί να έχουμε 4 12 εκατομμύρια σε ε, εξαγωγές, αλλά στην παρούσα κατάσταση αρκούν συν οι επιπτώσεις που υπάρχουν. Όλα αυτά δεν είναι αμεληταία. Δεν έχουμε όλα τα στοιχεία στα χέρια μας. Αυτό όσον αφορά τον ορισμό. Υπήρξαν δυσκολίες, όπως σας είπα, κατόπιν όμως υπάρχει και το πρόβλημα ε, των πολιτικών θεμάτων. Δεν υπάρχουν κριτήρια που θα ε, μας, ε, μας επιτρέψουν να πείσουμε χώρες να αλλάξουν πολιτική. Αυτό είναι γεγονός ότι πρέπει να παραμένουμε ανοιχτοί και προς το παρόν δεν είμαστε σε θέση να ασκήσουμε πίεση εφόσον δεν υπάρχει κοινή εμπορική πολιτική. Δεύτερη παρατήρηση, την οποία θα βρείτε πάλι σε μελέτη μας, είναι το θέμα του retaliation. Δεν μπορούμε να το ποσοτικοποιήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι σε τόσες περιπτώσεις θα έχουμε αντίπεινα, αντίμετρα. Αυτό πρέπει να το δούμε διαφορετικά και όχι μόνο από πολιτική άποψη. Ε, υπάρχει θεωρία ότι αν θεωρήσουμε ότι άλλες χώρες ε, κλείνουν συστηματικά, υπάρχει ε, μία προτίμηση όπως κάνει η τουρκική κυβέρνηση για την Αμερική πούμε, και την Ινδία. Ε, ε, τι κάνουν λοιπόν, επιβάλλουν εθνικούς κανόνες και αν αυτές οι χώρες με βάση αυτά τα πραγματικά γεγονότα λένε ότι θα λάβουν αντίμετρα επειδή με αυτόν τον τρόπο μπορούν ε, να διαπραγματευτούν με βάση την αμοιβαιότητα, αυτό δεν είναι παρά μία υπόθεση. Εκείνο το οποίο δεν περιλαμβάνει σε μελέτη αντικτύπου είναι ότι κανένας δεν μας είπε ότι αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη, ότι δεν υπάρχουν πλέον εμπορικές ανταλλαγές. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε τι συμβαίνει και να εξακολουθούμε να διαπραγματευόμαστε με την ελπίδα ότι θα προχωρήσουν τα πράγματα. Και πρέπει να σας πω ότι στις διαπραγματεύσεις, στι ε, στις συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, η Επιτροπή έχει προχωρήσει αλλά δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα επόμενα στάδια. Στη μελέτη αντικτύπου υπάρχει ένα κεφάλαιο που εξηγεί πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή, αυτή την έλλειψη μόχλευσης και να δούμε τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα και από πλευράς εμπορικών διαπραγματεύσεων. Επόμενο θέμα. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει ε, στην, στην εσωτερική αγορά. Η Επιτροπή διαιρεί την αγορά. Ε, υπάρχει αποκεντρωμένος μηχανισμός το ζητούμενο είναι κατά πόσον μπορεί αυτό να λειτουργήσει επειδή υπάρχουν οι κανόνες καταγωγής, η αλυσίδα τροφοδοσίας, η οποία είναι πολύ περίπλοκη. Αυτά όλα τα εξετάσαμε. Για παράδειγμα, για τους κανόνες καταγωγής, ε, σε ορισμένε περιπτώσεις, ε, οι προσφορές είναι θεμητέ, αυτό γίνεται και πιστεύουμε ότι οι επιχειρήσεις που έχουν αλυσίδα εφοδιασμού λειτουργούν σωστά, αλλά μερικέ φορέ οι επιχειρήσει βρίσκουν αυτό το σύστημα περίπλοκο. Απ' την άλλη πλευρά όμω, ο τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι λυσίδε εφοδιασμού και οι προμηθευτέ του είναι ικανοί, ε, αν θέλουν οι επιχειρήσει μπορούν να αλλάξουν προμηθευτή αν το επιθυμούν. Βεβαίω υπάρχουν ορισμένε ε, περιπτώσεις όπου το επίπεδο είναι πολύ ψηλό, που το όριο είναι πολύ ψηλό. Σκεφτήκαμε λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχει ένα όριο για τους κανόνες καταγωγής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πιστεύουμε. Κυρίως επειδή οι εταιρείε ε, με τις οποίες συζητήσαμε ε, το κάνουν για να υπάρχει πρόσβαση στις αγορές οι επιχειρήσεις δεν είπαν όλες μαζί ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν υπάρχει, ορισμένες, σε ορισμένε περιπτώσει είχαν ενδιασμού, αλλά δεν υπάρχει μια γενική τοποθέτηση. Επίση, εξετάσαμε την επιλογή των εμποδίων. Οι ενδιαφερόμενοι δεν συμφωνούν απόλυτα. Είναι κάτι το οποίο η Επιτροπή ε, δεν θα δεχόταν, διότι αν είχαμε καταλήξει σε ακραίε λύσει, δηλαδή είτε να κλείσουμε εντελώ την αγορά, είτε να γίνουν επιλεκτικέ διαπραγματεύσει. Εκείνο το οποίο θέλουν οι ενδιαφερόμενοι την πρώτη επιλογή, δηλαδή τον αμερικανικό τύπο. Δεν συμφωνούσαμε, πιστεύουμε, ότι ένας μηχανισμός ο οποίος διατηρεί ανοιχτή την αγορά πέραν των 5 εκατομμυρίων δεν είναι κάτι το οποίο ε, είναι δεκτό. Δεν κλείνουμε την αγορά για τις μεγάλες συμβάσεις, μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά τίποτα δεν γίνεται αυτομάτως. Και η εμπορική πολιτική θα εξασφαλίσει ότι ε, ε, αυτό θα αντιμετωπιστεί. Δηλαδή δεν μπορεί η δεξιά μας να κάνει κάτι, και η αριστερά μας να κάνει κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τις απόψεις στην εσωτερική αγορά και άκουσα τα θετικά σας σχόλια για την ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου οργάνου και θα σας εξηγήσω χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες το σκεπτικό πίσω από, αυτήν την, από αυτό το αποκεντρωμένο μέσο. Καταρχάς να σας υπενθυμίσω ότι Σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 10, το σκεπτικό είναι η δημιουργία αυτού του μέσου, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει μέτρα για να επιβάλλει ρυθμίσεις εάν υπάρχουν ορισμένα ε, προβλήματα ε, δομικά και διαρθρωτικά στην αγορά και αν υπάρχουν προβλήματα συνένεσης και συμφωνίας όσον αφορά την προσέγγιση. Καταρχάς, το σκεπτικό πίσω από αυτό το μέσο είναι η ρύθμιση των καθημερινών ε, δημοσίων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι που δεν ίσχυε πριν. Δεν μπορούσαμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στην αγορά στο παρελθόν σε αυτόν τον τομέα. Καταρχάς, δεν θα έπρεπε να επιβάλλουμε υποχρέωση να δέχονται οι αρχές ε, να αναθέτουν συμβάσεις από οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Αυτό που θέλουμε να δημιουργήσουμε στην περίπτωση αυτή είναι μια γκρίζα ζώνη για τις χώρες που έχουν την επιθυμία να ε, αναλάβουν μια σύμβαση. Έπειτα, η δημιουργία του οργάνου αυτού δεν επιβάλλει καμία απαργόρευση, όπως είπα. Δημιουργούμε μια γκρίζα ζώνη όσον αφορά τα νομικά δικαιώματα συμμετοχής σε προσφορές. Κατανοούμε ότι ως απορία αυτού του κανόνα το ερώτημα προκύπτει είναι ποιος θα είναι ο βασικός ο αρχικός κανόνας. Έχουμε αρχίσει την επεξεργασία της πρότασης αυτής και κατά βάση στόχος είναι η πρόσβαση στην αγορά σε τρίτες χώρες, ιδιαίτερα για συμβάσεις που γίνονται σε ευρώ. Οι συμβάσεις που ξεπερνούν το όριο των εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση το άρθρο 6 προβλέπει ότι υπάρχουν ξεκάθαρες προδιαγραφές που μπορούν να εφαρμοστούν εάν θέλουμε να αποκλείσουμε κάποιες τέτοιες ώρες. Καταρχάς πρέπει να υπάρχει έλλειψη αμοιβαιότητα από τις ε, χώρες αυτές για να τις αποκλείσουμε. Μετά, εάν υπάρχει πρόσβαση από ε, ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις σε αυτές τις χώρες που μπορούν να κάνουν προσφορά. Και σε περίπτωση που, ε, ένα, που μια χώρα θέλει να αποκλείσει ξένους επενδυτές, πρέπει να το κάνει αυτό βάσει κάποιων κανόνων που θα πρέπει να πληρούνται. Για τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι το άρθρο 6 συνεισφέρει σημαντικά και δημιουργεί τη δυνατότητα καλύτερης διαπραγματευτικής δύναμης, δυνατότητα μόχλευσης. Υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες που τίθενται όσον αφορά την αμοιβαιότητα και ένα ρυθμιστικό όργανο που θα φροντίζει να μην λαμβάνονται αυθαίρετες και επισφαλείς αποφάσεις. Εάν κάποια πόλη, κάποια περιφέρεια, παρόλα αυτά, θέλει να κάνει μια εμπορική συναλλαγή με χώρε με τι οποίε δεν υπάρχει συμφωνία, θα μπορεί να το κάνει, αλλά υπό ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Άκουσα τι ερωτήσει από, αυτές τις, από την Επιτροπή σα σχετικά με την εφαρμογή του μέσου αυτού. Θέλουμε να βρούμε λύση για τα προβλήματα που θίξατε και γι' αυτό είμαστε ανοιχτοί στη συνεργασία και τις προτάσεις σας. Ε, μπορούμε να βελτιώσουμε, πιστεύουμε, την πρόταση με τη συμβολή σας. Όμως πιστεύουμε πως παρόλα αυτά ένα άρθρο όπως το άρθρο 6 είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Πιστεύω πως τώρα είναι κατάλληλη στιγμή να ανοίξουμε τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή. Ποιος θα ήθελε λοιπόν να απευθύνει ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διευκρινήσεις, αποσαφηνήσεις σχετικά με την παρουσίασή τους. Για να εξαντώ. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία, όπως τα κοινωνικά θέματα, για παράδειγμα, που είναι πολύ σημαντικά εκεί η μόνη δυνατότητα περιορισμών προέρχεται από μία μη αμοιβαιότητα. Ούτε τα κοινωνικά θέματα, ούτε οι κρατικές προμήθειες υπησέρχονται στα κριτήρια που επιτρέπουν περιορισμούς. Πώς μπορείτε να δικαιολογήσετε ένα τέτοιο περιορισμό, αυτά τα όρια δηλαδή, στα κριτήρια που χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, πιστεύω ότι αναφερθήκατε στις ε, συνεχιζόμενες συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διεξάγονται. Στις συζητήσεις αυτές, οι κοινωνικές προμήθειες και οι πράσινες προμήθειες βρίσκονται σε πρώτη θέση. Να σας το τονίσουμε αυτό πριν τους σας ενημερώσουμε για το νέο καθεστώς. Υπάρχει μια ναι, διεθνή πολιτική, η οποία φυσικά θα ακολουθεί τους κανόνες που ε, έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτό το όργανο δεν θα ασχολείται με αυτού του τύπου της ερωτήσεις, διότι οι κανόνες θα υπάρχουν στις οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις. Υπάρχει τώρα άρθρο 7 της πρότασης και στο άρθρο αυτό θα δείτε ότι θα υπάρχει η ευκαιρία σε όσους κάνουν προσφορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποβάλουν προσφορά και να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός, θα υπάρχει δυνατότητα απόρριψης και θα υπάρχουν αναφορές στην κοινωνική διάσταση και σε κανόνες που πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Δηλαδή σε περίπτωση που θα έχουμε μία πολύ χαμηλή προσφορά θα υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο και θα τίθεται ε, κάποια κριτήρια, κάποια κοινωνικά κριτήρια επίσης. Μάλιστα. Ας κλείσουμε αυτήν την δεύτερη ανταλλαγή απόψεων και ας ακούσουμε τον εισηγητή κύριο Κάσπαρη. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ πολύ και την Επιτροπή. Ανυπομονώ να έρθει ο Φεβρουάριος και να μπορέσουμε να ασχοληθούμε περαιτέρω με την έκθεση αυτή. Επόμενο θέμα. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε το Φεβρουάριο, θα έχουμε δημόσια ακρόαση και ανταλλαγή απόψεων, τρίτη ανταλλαγή απόψεων το Μάρτιο. Προχωράμε τώρα στο σημείο 11. Η εξωτερική πολιτική αερομεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια γνωμοδότηση από την Επιτροπή Μεταφορών που είναι η αρμόδια διότι φυσικά ασχολείται με τη σφαίρα μεταφορέ. Ο εισηγητή είναι ο Ρόμπερτ Στέρντι, είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων και έχει Ρόμπερτ, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν ανέλαβα την υποχρέωση αυτή, πήρα μια ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είδα πόσο σοβαρή ήταν η υπόθεση αυτή σε επίπεδο νομοθετικό. Οι αερομεταφορές είναι βασικός συνεισφορέας της ευημερίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι η πρόσβασή μας μέσω των αερομεταφορών στις παγκόσμιες αγορές. Υπάρχουν πάρα πολλά πλέον εκτήματα. Παρακαλώ, μπορείτε να μην συζητάτε στο βάθος της αίθουσας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Όχι μόνο παρέχει υπηρεσίε προ αυτού οι οποίοι πετούν ή εργάζονται στον τομέα, αλλά παρόλα αυτά είναι κινητήρα ε, οικονομικό ε, δραστηριοτήτων όπω ο τουρισμό και το εμπόριο. 7,8 εκατομμύρια θέσει εργασία ε, απασχολούνται σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, έχει ένα κύκλο εργασιών 478 δις. Αν οι ευρωπαϊκές αερομεταφορές ήταν κράτος μέλος, σε επίπεδο ΑΕΠ θα ήταν το 7ο στη σειρά. 23. By air, over 650 billion in 2010. Πρόκειται λοιπόν για μια χρήσιμη γενικά ανάλυση της κατάστασης και η πρόοδος που έχει σημειωθεί στις εξωτερικές πολιτικές αερομεταφορών από το 2005 είναι σημαντική. Υπάρχουν βέβαια και προβλήματα και προκλήσεις που αφορούν τον τομέα αυτό σε μια ανταγωνιστική γενικά θα έλεγα σε μια ανταγωνιστική ε, αγορά και είναι σαφές ότι όλα αυτά δείχνουν τη σημασία, πάση που έχει η συγκεκριμένη αυτή η δραστηριότητα. Πρέπει να υπάρξουν εγγυήσει λοιπόν και για τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών εταιριών σε ξένες αγορές. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις και δεν θα πρέπει να υπάρχουν διοικητικά πλαίσια τα οποία να μην είναι ιδιαίτερα διαφανή και να οδηγούν σε στρεβλώσεις της αγοράς. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η Ρωσική Ομοσπονδία απέτυχε στην εφαρμογή των διεθνών υποχρεώσεών της και στην, δεν σε εφάστηκε τη συμφωνία που υπέγραψε στο τέλος του 2011 σχετικά με τους κανόνες που αφορούν την υπέρπτυση της Σιβηρίας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε καλύτερα μέσα για την παρουσία μας στις αναδυόμενες οικονομίες. Για τα επόμενα χρόνια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι στις, μεγαλύτερες, στις εννέα μεγαλύτερες εν πάση περιπτώσει αναδυόμενες αγορές που αντιπροσωπεύουν το ίμιση του παγκοσμίου ΑΕΠ οι επιχειρήσεις μας θα έχουν την δυνατότητα να ε, δραστηριοποιούνται στις περιοχές των χωρών αυτών και στις αγορές τους. Πέντε από τις δέκα μεγαλύτερες κινέζικες πόλεις δεν συνδέονται με δυτικοευρωπαϊκά αεροδρόμια. Οι πόλεις αυτές ε, ξεπερνούν τα 30 εκατομμύρια κατοίκων. Είναι σαφές λοιπόν ότι υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό εδώ, εμπορικό, και είναι κάτι το οποίο θα μπορέσει να ενισχύσει και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σχόλια των σκιωδών ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα για τα θέματα στα οποία αναφέρθηκα. Ε, τις προτάσεις τους θα τις συμπεριλάβω και θα ακούσω επίσης προσεκτικά και τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά θα αποσταλούν όλα για μετάφραση στο τέλος της εβδομάδας. Αν θέλετε να προσθέσουμε κάτι παρακαλώ να το δώσετε στους συνεργάτες μου ή σε μένα σύντομα. Ευχαριστώ. Έμαθα πολλά από σας. Δεν ήξερα ότι είναι τόσο σημαντική η δραστηριότητα αυτή, λέει ο Πρόεδρος. Λοιπόν, θα ξεκινήσει η συζήτηση τώρα. Λάγκερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο εξηγητή. Όντως, εξεπλάγην κι εγώ ο τομέας των αερομεταφορών είναι αποφασιστικός για την οικονομία στην Ευρώπη. 200% του ΑΕΠ. Πάνω από 5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τον ε, τομέα των αερομεταφορών. Και η εμπορική του διάσταση είναι επίσης ιδιαίτερης σημασίας, διότι εκεί συνειδητοποιούμε ότι παρά το ότι ο τομέας των αερομεταφορών μεγαλώνει, οι ευρωπαϊκές αερογραμμές παρουσιάζουν ύφεση και αυτό πρέπει να το ανταλύσουμε. Γιατί συμβαίνει αυτό. Όπως ανέφερε και ο εισηγητής, υπάρχει πιστεύω αθέμητος ανταγωνισμός και κατακερματισμός του κλάδου. Και πιστεύω πως βασικό είναι να υπάρχει έλεγχος για αποφυγή του αθέμητου ανταγωνισμού και επίσης να δούμε πώς μπορούμε να δώσουμε ευρωπαϊκή χρειά στα σύμφωνα για τις αερομεταφορές. Πώς να, και πώς θα μπορέσουμε και στον ε, τομέα των αερομεταφορών να τον προσαρμόσουμε στα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ Ελπίζω να υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενεργήσουμε προς το συμφέρον του εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ένα υψηλό ποσοστό στο μερίδιο της παγκόσμιας αγοράς στον κλάδο των αερομεταφορών. Θα πρέπει επίσης ο τομέας αυτός να έχει συμμετοχή σε, σε ένα διεθνές εμπορικό σύμφωνο Βλέπετε για παράδειγμα τι συμβαίνει με χώρες του ΟΣΑ όπως ο Καναδάς ή οι Ηνωμένε Πολιτείε. Εκεί πρέπει να δώσουμε βάση. Επίσης πρέπει και εμείς να πάμε διαβασμένοι διότι το θέμα του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού και η εφαρμογή του δεν είναι, έχει ακόμα λυθεί. Είναι ακόμα ανοιχτό. Επίσης η χωρητικότητα είναι και αυτό ένα θέμα που παραμένει ανοιχτό. Και επίση, τα κοινωνικά στάνταρ και τα περιβαλλοντικά στάνταρ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θέμα που πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το συνδέσουμε ιδιαίτερα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Πρέπει και αυτά να ληφθούν σοβαρά υπόψη στο σύμφωνο για τις αερομεταφορές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πολύ ευτυχής που μπορούμε ακόμα να υποφεληθούμε τον Ρόμπερτο Νίκ, τον ε, Βρετανό Ευρωβουλευτή. Υπάρχει μία διάσταση που ο εισηγητής ε, δεν ανέφερε επί της οποίας η Επιτροπή δεν επιμένει πολύ. Φαντάζομαι ότι ε, αυτό είναι το θέμα του κλίματος στην ευρωπαϊκή επικαιρότητα υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο, δηλαδή η βούληση να υποβληθεί η αεροπορία στην κοινή πρακτική, δηλαδή ε, στην αγορά ποσοστώσεων, του άνθρακος, που υποστηρίζει και όλο το Κοινοβούλιο. Σε αυτό το σύστημα λοιπόν, και ακόμα όταν συζητάμε με τους συμπολίτε μας, πάντοτε δεν καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι όταν παίρνουν το αυτοκίνητό τους να πάνε στη δουλειά πληρώνουν σημαντικούς φόρους και όταν πάρουν το αεροπλάνο είτε για το δίκτυο του άνθρακα όπως για την κυροζήνη δεν πληρώνουν φόρους είχε γίνει μια διαπραγμάτευση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αεροσυπλοεία και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή και είχαμε συμφωνήσει, είχαμε καταλήξει μια συμφωνία η οποία φαινόταν έξυπνη για όλους. Και μετά έγιναν λόμπις από πολλές αναδυόμενες χώρες και ξαφνικά η Κομισιόν αποφάσισε να αναστείλει κατά κάποιο τρόπο αυτόν τον κανονισμό και να παραπέμψει αυτό σε διεθνές επίπεδο. Υποστηρίζουμε έντονα την ιδέα μιας συμφωνίας, κυρίως στα πλαίσια ε, του ΙΚΑΟ, και να έχουμε ένα ε, παγκόσμιο σύστημα που να αφορά τις αερομεταφορές. Και αυτό είναι από τα στοιχεία των διαπραγματεύσεων. Αλλά νομίζω ότι εδώ η Ευρώπη είναι αρκετά σημαντική ήπειρος από πλευράς των αερομεταφορών. Προκειμένου αυτή η Ευρώπη να μπορεί να αναλάβει την ηγεσία σε αυτό το τομέα. Και οι αερομεταφορές είναι ένας τομέας ε, που έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά τι εκπομπέ του άνθρακο. Διπλασιάστηκαν οι εκπομπέ αυτέ από το 1970. Αυτό έχει τονιστεί. Είναι ένα αναπτυσσόμενο κλάδο. Συνεπώ πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό ο παράγον του κλίματο, ε, του θορύβου να ληφθούν υπόψη ώστε να έχουμε μια ηγετική θέση στην Ευρώπη ώστε ε, να ε, γνωρίσουμε ποιος είναι ο ρόλος, σημαντικός ρόλος των αερομεταφορών. Άλλα ερωτήματα. Κυρία Βέρνερ. Κυρία Βέρνερ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη. Πολύ θετικά λόγια άκουσα για την ανακοίνωση αλλά και για την σημασία του τομέα των αερομεταφορών στην ευρωπαϊκή οικονομία. Οι αερομεταφορές στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν κρίση. Και όχι μόνο, όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει κρίση. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που κάναμε αυτή την ανακοίνωση. Έγινε η αναθεώρηση της πολιτικής ε, για τις αερομεταφορές και μετά από Εκτενής διαβουλεύσεις το Σεπτέμβριο αποφασίσαμε να συμπέσουμε και με την δέκατη επέτειο της πολιτικής για τις αερομεταφορές, διότι το 2002 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξεδώσε την απόφαση για τον Ευρωπαϊκό Ουρανό. Γεγονός είναι ότι έχουμε μεγάλα αεροδρόμια, μεγάλη βιομηχανία αερομεταφορών. Το ΑΕΠ είναι μεγάλο, όπως είπε και ο εισηγητής. Δεν πρέπει όμως να το θεωρούμε αυτό δεδομένο. Πρέπει να προσπαθήσουμε, και αυτό το τονίζουμε και στην ανακοίνωση, να τονίσουμε όχι μόνο τα επιτεύγματα, αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε για να διατηρήσουμε τη θέση στην οποία έχουμε βρεθεί. Ε, ένα ζήτημα φυσικά είναι ο κατακαιρματισμός, ο εθνικός, ο οποίος επιμένει, η έλλειψη ε, αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό που χρειαζόμαστε πραγματικά είναι μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή διάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με χαρά της έλαβε θετικά σχόλια και συμπεράσματα για την ανακοίνωση. Φυσικά και θα μπορούσαμε να είμαστε πιο φιλόδοξοι στην κατάρτιση της ανακοίνωσης. Όσον αφορά το περιβαλλοντικό ζήτημα και τη διάσταση στον τομέα των αερομεταφορών, θα ήθελα να πω ότι υποστηρίζω απόλυτα την συνεχιζόμενη προσπάθεια να λυθεί το θέμα σε παγκόσμιο επίπεδο και να δοθούν εγγυήσεις για θεμητό ανταγωνισμό στον τομέα των αερομεταφορών στην Ευρώπη. Αυτό που θέλουμε να δούμε εμείς στην έκθεση είναι να υπάρξει μια δυνατότητας ευελιξίας. Ο εισηγητής ανέφερε την κατάσταση με τις αναδυόμενες αγορές και να τονίσω επίσης τις δυνατότητες να προασπίσουμε καλύτερα τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών ε, εταιριών και της βιομηχανίας έναντι στον αθέμητο ανταγωνισμό. Έτσι ώστε να έχουμε και δυνατότερη διαπραγματευτική θέση. Πολλές φορές ε, έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολους εταίρους. Σε γενικές γραμμές, η αναθεώρηση του μέσου προγραμματίζεται για το 2014. Εκρεμούν και εξελίσσονται αυτή τη στιγμή αρκετές διαπραγματεύσεις και υπάρχουν αρκετές χώρες οι οποίες θέλουν να εισέλθουν σε συμφωνίες το στομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για να κλείσουμε αυτήν την διαβούλευση, ας δώσουμε ξανά το λόγο στον εισηγητή κύριο Στέρντι. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννικ. Προσπαθώ να είμαι σύντομο όταν κάνω μια έκθεση και έπρεπε να αφήσω κάτι απ' έξω, έτσι ώστε να έχει και εσύ κάτι να πει. Έχει απόλυτο δίκιο. Το παραλείψαμε. Το είχα υπόψη μου, βέβαια. Αλλά να πω ότι όταν έχουμε εργαστεί ένα χρόνο πάνω σε αυτό, όταν υπάρχει προηγούμενο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τότε θα μας πει ότι έχουμε περιθώριο opt-out για ένα χρόνο, έχει επιπλοκές αυτό το ζήτημα, διότι τότε ενδεχομένως μπορεί να υπάρξουν εταιρείε που δεν θα θέλουν να αγοράσουν ένα ευρωπαϊκό αεροσκάφος, για παράδειγμα. Μπέντ, θα συνεργαστούμε στενά, διότι έχουμε τις ίδιες απόψεις και είμαστε και στην Επιτροπή Μεταφορών. Είναι πραγματικά συναρπαστικό, διότι αυτή η έκθεση είναι μια έκθεση στην ε, οποία βλέπουμε τόσες ενδιαφέρουσες απόψεις και όταν άρχισα να διαβάζω το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό είναι για την Ευρώπη και για τις θέσεις εργασίας και για την οικονομία μας. Πόσο, πόσοι μας είπατε απασχολούνται 7 εκατομμύρια στον τομέα των αερομεταφορών. Πρέπει να μην κάνουμε κανένα λάθος λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντα και κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να μα ενημερώσετε και για το χρονοδιάγραμμα έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μα και να γίνουν και οι μεταφράσει για τι τροπολογίε. Βεβαίω. Η επόμενη συνεδρίασή μας, τον Φεβρουάριο, εκεί θα συζητήσουμε τις ε, τροπολογίες. Το Μάρτιο θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή τον Μάρτιο επίσης. Έχουμε δύο μήνες, δηλαδή. Να τονίσω κι εγώ, να υπογραμμίσω τη σημασία της γνωμοδότησης αυτής. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα. Εμπορικά. Όχι και όχι μόνο. Ναι, η Βρετανία ακόμα δεν μας έχει εγκαταλείψει. 2017-2018 τότε ίσως. Η ανακοίνωση του κυρίου Κάμερος είχε ως εξή. το 2015 υποσχέθηκε στους Βρετανικούς ψηφοφόρους να διεξάγει δημοψήφισμα για το αν θα παραμείνουν ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Σημείο 15 τώρα. Και αυτό πολύ σημαντικό. Αφορά το ποιος θα έχει την οικονομική ευθύνη σε περίπτωση διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών που προβλέπονται από διεθνείς συμφωνίες, στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλόμενο μέρος. Μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν αυτό, έχουν το δικαίωμα πρωτοβουλίας. Ο δικός μας εισηγητής είναι ο Παύλ Ζαβέλσκι, Ζαλεύσκι. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων σήμερα και ανυπομονούμε να σας ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε αυτό το σχέδιο κανονισμού είναι η φυσική συνέχεια της προηγούμενης και δεν είναι λιγότερο ο κανονισμός δεδομένου ότι επηρεάζει τον, τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη όσον αφορά τις πληρωμές που έχουν σχέση με την ε, οικονομική ευθύνη μετά από τις δυτικές αποφάσεις. Αυτό βασίζεται στο σωστό πλημερισμό της οικονομικής ευθύνης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους μέλους του. Αλλά το βασικό πρόβλημα είναι πώς να προβλέψει κανείς όλα τα πιθανά σενάρια περιπτώσεων ε, που έχει ο εναγόμενος και πώς θα γίνει η τελική κατανομή του οικονομικού βάρους να αφορά την υποχρέωση να κατευθυνθούν τα βάρη. Η... Είναι ισορροπημένη η έκθεση της Επιτροπής και αποτελεί μια καλή βάση για συζητήσεις και για την εκπόνηση της τελικής εκδοχής που μπορεί να υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αλλά περιέχει ορισμένες διατάξεις που δεν είναι αρκετά σαφείς ε, και χρειάζεται να διευκρινιστούν. Αυτά τα θέματα λοιπόν είναι τα βασικά στοιχεία της έκθεσής μου. Συνοψίζοντας, ο συλλογισμός ε, των τροπολογιών που προτείνω είναι ο εξής. Αφορά τα εξής θέματα. Θα ήθελα να επιφέρω ορισμένε αλλαγέ στο άρθρο 2 το οποίο αφορά τους ορισμούς. Πιστεύω επίσης ότι μπορούμε να ορίσουμε καλύτερα τη λέξη μεταχείριση, treatment, που χρησιμοποιείται πολλές φορές από τον κανονισμό. Αλλά δεν έχει οριστεί στην πρόταση της Επιστροπής. Κατόπιν θα ήθελα να διευκρινίσω ορισμένα τμήματα του άρθρου 8.2 και του άρθρου 9.2, ώστε να, είναι, να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια, ορίζοντας ποιος είναι ο συλλογισμός επιτροπής ε, πίσω από το αίτημα που ζητεί να αναλάβει την περίπτωση ή να ζητήσει από ένα κράτος μέλος ε, να τοποθετηθεί με κάποιο τρόπο. Θα πρέπει εδώ να υπάρχει ένα συμφέρον της κοινότητας που αδιαπνισβήτητα διακυβεύεται. Στο άρθρο 33 δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το επίπεδο της οικονομικής ευθύνης του των κρατών μελών όταν αυτή η διάταξη έχει εφαρμογή. Κατόπιν, όπως είπα πρωτήτερα, έχω επιφυλάξει σχετικά με τη διατύπωση του άρθρου 18.1 σχετικά με τις προκατεβολές ε, των δαπανών διατησίας. Το ερώτημα είναι ε, ε, τι αντίκτυπο έχει αυτός, αυτή η διάταξη, λαμβάνοντας υπόψη πολλές διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών. Στο άρθρο τώρα 21 προτείνω περισσότερες λεπτομέρειες, πιο λεπτομερή περιγραφή σχετικά με την υποχρέωση Επιτροπής να δώσει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Νομίζω ότι πρέπει να καθορίσουμε ε, τι είδους πληροφορίες αναμένουμε από την Επιτροπή. Για παράδειγμα, πιστεύω ότι θα πρέπει να ενημερωθούμε επίσης σχετικά με τις περιπτώσεις, τη διατησίας και τα αποτελέσματα που έχουν επειδή πιστεύουμε όλοι ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη διαφάνεια. Κατόπιν, όταν μιλήσαμε με τους σκιώδους ηγητές, πολλοί συνάδελφοι είχαν τη γνώμη, και εγώ το πιστεύω, σχετικά με αυτό τον όρο regulation, κανονισμός, αλλά οι ίδιες οι συνθήκες στις, όσον εδώ περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει, μισχωρείτε, στις περιπτώσεις, περιπτώσεις θα πρέπει να αποφεύγουμε διαιτητικές διαδικασίες και απλά και μόνον να αναφερόμαστε στις νομικές διαδικασίες που προβλέπονται. Σε αυτές τις χώρες όπου το κράτος δικαίου εφαρμόζεται σωστά. Αυτά, αυτές είναι οι πρώτες παρατηρήσεις μας ε, για να ξεκινήσει η συζήτηση και θα ήθελα να ακούσω την άποψη και των άλλων συναδέλφων και της Επιτροπής ώστε να μας βοηθήσουν σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Ζαλέσκη. Υπάρχει δυνατότητα δηλαδή για τροπολόγηση των προτάσεων της ε, Επιτροπής. Ε, αυτά που μας είπατε δείχνουν ότι γενικά συμφωνείτε με την πρόταση της Επιτροπής. Πράγματι έχει σημασία ο φάκελος αυτός. Το είχαμε προτείνει εμείς στα πλαίσια της έκθεσης Καντέρ Αρίφ σχετικά με τις έμεσες, ε, άμεσες ξένες επενδύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται αρμοδία για τέτοιου είδους διεθνείς συμφωνίες που αφορούν τις άμεσες επενδύσεις. Και γι' αυτό απαιτείται να ρυθμίσουμε το θέμα της ευθύνη για τις ζημίες τις οποίες υφίστανται οι επενδυτές. Ας περάσουμε τώρα στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μιλώ εξ ονόματος του David Μάρτιν, του σκιώδους εισηγητή. Ο David Μάρτιν δεν μπορούσε να βρίσκεται μαζί μας σήμερα. Όντως, είναι αποφασιστική σημασίας πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με αυτό θα επιτευχθεί σαφήνεια. Και με την ενεργειακή χάρτα και με τα αναμενόμενα σύμφωνα με τον Καναδά βρισκόμαστε σε μια θέση όπου κοντεύουμε να φτάσουμε στο τέλος, δεν έχουμε ακόμα σαφείς κανόνες βέβαια. Από την άλλη, είπατε και εσείς, πρέπει να δούμε αν είναι αναγκαίο εδώ να δημιουργήσουμε μία νέα διαδικαστική ρύθμιση. Δεν ξέρω αν είναι αναγκαίο. Εάν αυτό είναι αναγκαίο να περιέχεται στο σύμφωνο και γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται να υπάρχουν σαφείς κανόνες. Και όπως είπε και ο εισηγητής, είναι εξαιρετικά σημαντική οι σαφείς κανόνες όσον αφορά την οικονομική ευθύνη ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω πως χρειαζόμαστε μια πολύ γρήγορη ρύθμιση και συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο. Ιδιαίτερα για το θέμα αυτό. Υπάρχει επίσης μια μεγάλη συμφωνία ανάμεσα στον Τέβιτ Μάρτιν και στον εισηγητή Γι' αυτό και θεωρούμε ότι η εργασία και η συνεργασία ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική. Κάποια σημεία θα ήθελα να τονίσω, τα οποία για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Ορισμένα τα ανέφερε και ο εισηγητής στις προτάσεις του. Αρχίζω με την μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν διαπραγματεύσεις οι οποίες δεν γίνονται ανοιχτά, γίνονται στα κρυφά, δεν ξέρουμε ποιος έχει την ευθύνη στο τέλος. Σίγουρα υπάρχουν εμπορικά ε, απόρριτα, όμως όσον είναι, όσο είναι δυνατόν πρέπει να εγγυηθούμε διαφάνεια. Έπειτα, όπως και είπε και ο εισηγητής, το ζήτημα του ρόλου του Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό. ή Ιδιαίτερα όσον αφορά την υποχρέωση σύνταξης εκθέσεων από το Κοινοβούλιο και προς το Συμβούλιο. Και αυτό πρέπει να το αναλύσουμε διεξοδικά και να δούμε την σχέση και την αναλογία των ε, πράξεων κατά εξουσιοδότηση και των εκτελεστικών πράξεων στον κανονισμό. Διότι είναι πολύ σημαντικό να αποφασίσουμε ποια είναι τα σωστά μέσα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Πιστεύουμε και εμείς όπως και ο εισηγητής ότι χρειάζονται ορισμένες γλωσσικές διευκρινήσεις και διευκρινήσεις στην διατύπωση έτσι ώστε να μην υπάρχουν τόσο μεγάλα περιθώρια ελιγμών. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στα συμφέροντα των κρατών μελών όταν υπάρχει ένα ζήτημα ιδιαίτερου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Δεν, ενδιαφέροντος. Δεν είναι όμως σαφές ποιο είναι αυτό το ζήτημα. Τι καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρον ένα θέμα. Αυτό χρειάζεται έναν καλύτερο και σαφέστερο ορισμό και περισσότερη σαφήνεια. Μετά το επόμενο σημείο που έχει μεγάλη προτεραιότητα για μας είναι του πού βρίσκονται τα όρια μεταξύ επίσημης και ανεπίσημης συμφωνίας. Εδώ πέρα πρέπει να δημιουργηθεί μια ξεκάθαρη ιεράρχηση, ώστε να εγγυηθεί και η μέγιστη δυνατή παροχή πληροφοριών σε περιπτώσεις ε, διαιτησίας. Αυτά προς το παρόν και να πω εκ μέρους του David Μάρτιν ότι χαίρεται για τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους των Πράσινων η Φραντσίσκα Κέλλερ, η οποία είναι επίσης και όδηση συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ζαλεύσκη. Ευχαριστώ και για την συνεργασία σας με εμάς τους και συγγετές που ήταν πολύ χρήσιμη. Συμμεριζόμαστε τις αμφιβολίες και τις ανησυχίες τις οποίες αναφέρθηκατε Νομίζω ότι τα δικαστικά συστήματα μπορούν να δώσουν ε, δίκαιες μορφές διαιτησίας και γι' αυτό οι επενδυτές δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο και πιο ευνοϊκά από τους εθνικούς επενδυτές. γιατί οι εθνικοί επενδυτές δεν έχουν τη δυνατότητα να στραφούν σε διεθνή επίπεδα διατησίας. Ξέρουμε τώρα περιπτώσεις εις βάρος χωρών όπως ε, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία, όπου εκεί υπάρχει μια, δημιουργείται μια διαφορετική αντιμετώπιση ανάμεσα στις δύο κατηγορίες επενδυτών, ξένους και εθνικούς. Αυτό είναι άδικο, πρέπει να αντιμετωπιστεί και οι υπόλοιπε χώρες του ΩΣΑ θα πρέπει να προσπαθήσουν να καλύψουν τις, τα κενά τα οποία υπάρχουν έτσι ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι τους οποίους διατρέχουν οι επιχειρήσεις. Δεν θα αρχίσω εδώ να σχολιάσω τα υπέρ και τα κατά του ISDS, αλλά παρόλα αυτά το Κοινοβούλιο έτσι και αλλιώς δεν είχε τη δυνατότητα να εκφραστεί από αυτού. Και ναι μεν οι επενδύσεις είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουμε κανένα λόγο σε αυτήν. και θα πρέπει η γνωμοδότηση να μας δώσει μια, η Επιτροπή μάλλον να μας δώσει μια γνωμοδότηση σχετικά με τα διάφορα επίπεδα τα οποία θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Το θέμα είναι ότι το ISDS δίνει την δυνατότητα σε διεθνή δικαστήρια να κρίνουν για την καταλληλότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τη συμβατότητά της με τα εθνικά δικαϊκά συστήματα και νομίζω ότι αυτό όπως και η νομολογία των διεθνών δικαστηρίων γύρω από τα θέματα τα επενδυτικά μπορεί να δημιουργήσει σε νέες καταστάσεις αβέβαιες. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι αν οι νομικές ρυθμίσεις που προκρίνουμε εμείς αυτό εδώ το κοινοβούλιο μπορεί να αμφισβητηθούν ή όχι από διεθνείς ε, επενδυτές και αν θα χρησιμοποιηθούν τέτοιες διαδικασίες υπέρ της καταχρηστικής, αν θέλετε, προσκόμισης αποζημιώσεων. Έχει συμβεί στο παρελθόν αυτό. Ξέρετε ότι υπάρχει μια ολόκληρη γενιά επενδυτικών νομικών οι οποίοι αναζητούν απασχόληση και θα εκμεταλλευτούν τα συστήματα αυτά. Υποστηρίζουμε την τελευταία παρατήρηση που έκανε ο εισηγητής και ελπίζουμε ότι στην έκθεσή σας θα καλύψετε αυτά τα κενά και τις ανησυχίες μας σχετικά με τους μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των διλημάτων αυτών. Ίσως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να μπορούσε να αποκτήσει κάποιο ρόλο εδώ, ελέγχοντας το αποδεκτό ημί τέτοιων περιπτώσεων. Και εφόσον κρυθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι δεν είναι αποδεκτή μια τέτοια προσφυγή, ε, θα μπορεί ο προσφεύγων να επιστρέψει στα εσωτερικά δικαστήρια ή στην διεθνή σφαιρικά γενικότερα διατησία. Δεν πρέπει να δημιουργούμε λοιπόν εμείς ε, ένα επιπλέον επίπεδο απονομής δικαιοσύνης, αλλά να προσπαθήσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες ε, του επενδυτή και την προσπάθειά του να δικαιωθεί. Νομίζουμε λοιπόν ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα ήταν χρήσιμος για να εκφράσουμε κάποιες μορφές αιρεσιμότητα σε ορισμένα από τα θέματα τα οποία, στα οποία αναφέρεται το ISDS και νομίζω ότι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμεριζόμαστε τις ίδιες ανησυχίες. Καλώς σας ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. η εκπρόσωπος της Επιτροπής είναι τακτική θαμών της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Ζαλέτσκι και τους σκιώδεις εισηγητές για τα σχόλιά τους και την εισαγωγή τους σήμερα. Κάποιες γενικές εισαγωγικές παρατηρήσεις και μετά να αναφερθώ σε τρία θέματα στα οποία έγιναν ήδη αναφορές σήμερα. Καταρχά, θα πρέπει να πάμε λίγο προς τα πίσω και να δούμε ακριβώς το θέμα των αρμοδιοτήτων και ποιο είναι ο στόχος και η εμβέλεια της συγκεκριμένη πρότασης. Δεύτερον, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα ειδικά θέματα που θέτουν τα μέλη του Κοινοβουλίου. Και τρίτον, ένα σχόλιο για κάποιες από τις ερωτήσεις οι οποίες στέθηκαν σχετικά με το καθεστώς των επενδυτών τα μέλη έθεσαν ερωτήσεις που ίσως να μην είναι και το αντικείμενο της σημερινής συζήτησης, αλλά εφόσον μπορεί, εφόσον είναι δυνατόν, μπορούμε να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις για τις δυνατότητες που υπάρχουν να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες αυτές. Όπως είπατε, ο κανονισμός αυτός είναι ένα απαραίτητο σύνολο προτάσεων για να καλυφθεί ένα κενό το οποίο ε, έχει δημιουργηθεί με τις νέες αρμοδιότητες για το τομέα των επενδύσεων που ε, ήρθαν στην επικαιρότητα μέσω του άρθρου του 7 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Προσπαθούμε λοιπόν εμείς να δείξουμε ότι όταν τεθούν σε συμφωνία οι επενδυτικές ευρωπαϊκές συμφωνίες θα υπάρχει απόλυτη νομική ασφάλεια σε σχέση με αυτές. Αυτή είναι η πρότασή μας. Το πρώτο θέμα αφορά, όπως είπα, τις αρμοδιότητες και τη δικαιοδοσία, επαναλαμβάνω, ότι επί της ουσίας σύμφωνα με το 2007 έχουμε την αρμοδιότητα σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση της εξωτερικής αντιπρόσωπησης. Αυτό δεν είναι κάτι το καινούργιο επιβεβαιώθηκε επανειλημμένα τις τελευταίες δεκαετίες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και αυτό ισχύει επίσης και στις επενδύσεις όπως αυτές καλύπτονται από το 2007 της συνθήκης. Έχουμε πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας σε σχέση με τον ΠΟΕ στην Επιτροπή στα πλαίσια της εκπροσώπησης των συμφέροντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντίστοιχες τέτοιες νομικές αρχές εφαρμόζονται και στη δική μας περίπτωση. Όμως, Το θέμα της ρύθμισης των διαφορών για τους επενδυτές, ναι μεν περιλαμβάνεται στην εξωτερική αντιπροσώπευση τη δική μας, όλα αυτά υπάρχουν ορισμένες πλευρές που αφορούν τις ε, ρυθμίσεις, αν θέλετε, των ε, διαφορών για τους ε, επενδυτές που απαιτούν κάποια μέσα πιο συγκεκριμένα, πιο κατάλληλα μέτρα τα οποία να είναι ευθυγραμμισμένα με τα ειδικά χαρακτηριστικά των περιπτώσεων για τις οποίες υπάρχουν διαφορές. Ως εκ τούτου λοιπόν στην πρότασή μας εμείς λέμε ότι ο κανόνας ο οποίος μπορεί να αλλάξει, το default rule εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μια επιπλέον αρμοδιότητα, και η δυνατότητα αντιπροσώπευσης στη συγκεκριμένη περίπτωση ακολουθεί την πράξη η οποία βρίσκεται υπό αμφισβήτηση από πλευρά των επενδυτών. Δηλαδή δεχόμαστε μια εξαίρεση στο γενικό κανόνα της εξωτερικής αντιπροσώπευσης. Ε, η εξαίρεση αυτή, επαναλαμβάνω, πρόκειται για μια πολύ σημαντική εξαίρεση και είναι κάτι το οποίο έχει σχέση και συνδέεται, εν πάση περιπτώσει, με την πράξη, με τη σύμβαση η οποία βρίσκεται υπό αμφισβήτηση και αν στην ε, σύμβαση αυτή συμμετέχει ένα κράτος μέλος, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το κράτος μέλος ε, να εκπροσωπείται. Ταυτόχρονα η αρχή της ενότητας της εξωτερικής αντιπροσώπευσης όμως είναι κάτι το οποίο εδράζεται στο κοινό συμφέρον και θα πρέπει να διασφαλιστεί έτσι ώστε η χορηγούμενη εξαίρεση να είναι πλαισιωμένη σωστά σε νομικό κοινοτικό επίπεδο έτσι ώστε οι πράξεις ενός κράτους να μην δημιουργούν προβλήματα σε σχέση με τη συνολική κοινοτική αρμοδιότητα. Πρέπει λοιπόν να λαμβάνουμε πάντα υπόψη και το κοινοτικό συμφέρον. Αυτά λοιπόν στηρίζουν τον προτινόμενο κανονισμό που θα μας δώσει τη δυνατότητα εμάς στην Επιτροπή που δρούμε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιπροσωπεύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα όταν διακυβεύεται ένα κοινοτικό συμφέρον. Συμφωνούμε όλοι ότι είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε πως το κοινοτικό συμφέρον λαμβάνεται πλήρως υπόψη με έναν τρόπο ο οποίος να δίνει τη δυνατότητα επίλυσης διαφορών όποτε αναδύονται για επενδυτικές δραστηριότητες. Τώρα, για τα επιμέρους θέματα που έθεσαν οι βουλευτές. Υπήρξε ένα θέμα διαφάνειας σχετικά με το άρθρο 21. Θα ήθελα να πω ότι εμείς στο συγκεκριμένο θέμα έχουμε κάνει κάποια βήματα για να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας γύρω από τις ευρωπαϊκές συμφωνίες, περισσότερο από τις στις διμερείς επενδυτικές συμφωνίες. Έχουμε δώσει τη δυνατότητα ανοιχτών συνεδριάσεων σε αυτή την περίπτωση. Το κάνουμε και στις μεμονωμένες συμφωνίες, συμπεριλαμβάνοντας κάποιες ρήτρε διαφάνειας πιο σημαντικές και βαρύτερες από ό,τι στο παρελθόν και το κάνουμε επίσης και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της επικοινωνίας και της εμπλοκής μας με εσά και την Επιτροπή σας. Ένα μέλος του Κοινοβουλίου παρατήρησε ότι δεν υπήρξε εμπλοκή σε σχέση με το αρχικό κείμενο. Είναι αλήθεια, αλλά εγώ έχω έρθει σε αυτή τη συνεδρίαση στην Επιτροπή επανειλημμένα τον προηγούμενο χρόνο και και των θυρών και έφεσα ε, τις προθέσεις μας, παρουσίασα το κείμενο το ίδιο ε, και νομίζω αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Γιατί το πώς φαίνεται το κείμενο αυτό έχει σημασία και με μια ξεχωριστή νομική συζήτηση που μένει να γίνει. Λοιπόν, αυτά. Περιμένω συγκεκριμένες προτάσεις από πλευράς των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για περισσότερη διαφάνεια. Τέθηκε και άλλη μια ερώτηση σχετικά με τα θεσμικά διοργανικά θέματα, εφαρμοστικές πράξεις, πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Άρθρα 2.90 και 2.91. Νομίζω ότι έχουμε μια κοινή αντίληψη ερμηνεία των συγκεκριμένων άρθρων, αλλά θα επανέλθουμε στη συζήτηση. Τρίτον, αρκετά μέλη του Κοινοβουλίου έθεσαν τα θέματα των άρθρων 8 και 9. Και το θέμα του πιθανού ορίου ερμηνείας ή περιθωρίου ερμηνείας, το οποίο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την εφαρμογή των 8 και 9. Είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε εκ νέου ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα είναι σαφές στη συγκεκριμένη περίπτωση, ισχύει στην περίπτωσή μας, ισχύει η ενότητα της εξωτερικής αντιπροσώπευσης της Ένωσης και αυτό απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι σε θέση να εμπλακεί σε συζητήσεις, να κάνει προτάσεις, να μοιράζεται εμπειρίες και πληροφορίες. Εν σε αυτό βέβαια καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι σχετικά διακριτική σε σχέση με τις επικοινωνίες αυτές Έχουμε βρει μια σωστή ισορροπία ανάμεσα σε επαρκείς πληροφορίες που δίδονται από τη μία, που δημοσιοποιούνται από τη μία. Δημοσιοποιούμε τις περιπτώσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν γνωστές, αλλά και ταυτόχρονα προσπαθούμε να κρατήσουμε στην άκρη αυτά τα οποία δεν διευκολύνουν την εξέταση της υπόθεσης εάν δημοσιοποιηθούν. Είναι μια δύσκολη κρατησουμε στην ακρη αυτα τα οποια δεν διευκολυνουν την εξεταση της υπόθεση εαν δημοσιοποιηθουν ειναι μια δυσκολη ισορροπια σεβόμεθα πλήρως, προσπαθούμε να σεβαστούμε πλήρως την αρχή της ενότητας και της έκφρασης με ενιαίο τρόπο του κοινοτικού συμφέροντος. Υπήρξαν και κάποια άλλα σχόλια για το θέμα της ευκρίνειας του άρθρου 30, όχι του 13 συγγνώμη και του 18. Είναι τεχνικού τύπου άρθρα αυτά και μπορώ διμερώς να επικοινωνήσω με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν θέλετε, σε, ανεπίσημη, σε ανεπίσημο επίπεδο. Ένα τρίτο, μια τρίτη σειρά θεμάτων τώρα είναι εκτός κανονισμού. Είναι το εάν είναι απαραίτητη η δυνατότητα αυτή που δίδεται στους επενδυτές τα πλαίσια των διεθνών συμφωνιών όταν υπογράφονται συμβάσεων. Είναι απαραίτητο όταν διαπραγματευόμαστε μια τέτοια συμφωνία όπου υπάρχει κράτος δικαίου να υπάρξει μια τέτοια ρύθμιση. Λέμε ναι. Όταν επενδυτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνουν σε τρίτες αγορές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι χαίρουν της προστασίας που έχει γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευση σε κοινοτικό επίπεδο. Αν δεν συμπεριλάβουμε μια μέθοδο, μια διαδικασία προστασίας των συμφερόντων των επενδυτών, είναι σαφές ότι τα εσωτερικά, τα εθνικά δικαστήρια των χωρών αυτών δεν θα εφαρμόσουν τις ε, αποφάσεις ε, των ευρωπαϊκών δικαστηρίων ή τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Απαιτείται λοιπόν να διασφαλίσουμε υψηλό επίπεδο προστασίας για τους επενδυτές μα και ταυτόχρονα θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ότι η προστασία αυτή πρακτικά θα ληφθεί υπόψη σε περιπτώσεις διαιτησία, γιατί αλλιώς είναι κάτι το οποίο θα παραμείνει θεωρητικό. Είναι λοιπόν σε πολλές περιπτώσεις απαραίτητο να επιβληθεί η, αν θέλετε, η εφαρμογή αυτών των αρχών μέσω της διαιτησίας. Ε, αναφέρθηκα στο θέμα της διαφάνειας ε, προηγουμένως στα σχόλιά μου. Είναι κάτι το οποίο λαμβάνουμε πάρα πολύ σοβαρά και το οποίο θα θέλαμε να βελτιώσουμε σε επίπεδο συμφωνιών. Υπήρξε μια άλλη ερώτηση για την ισότιμη αντιμετώπιση των επενδυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν αφορά το θέμα των, της ρύθμισης των διαφορών, αλλά του είδους της προστασίας που προσφέρουμε εμείς στα πλαίσια των συμφωνιών των διεθνών. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι διασφαλίζεται μια κάποια ισορροπία ανάμεσα στις δύο κατηγορίες Αυτό είναι κάτι που μας απασχολεί, εν πάση περιπτώσει, όταν διαπραγματευόμεθα τέτοιου είδους συμφωνίες, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ανήκει στο θέμα της επίλυσης των διαφορών, είναι κάτι το οποίο αφορά γενικότερα την προστασία των επενδυτών και στο εσωτερικό θεσμικό πλαίσιο και εδώ τίθεται και το θέμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τις σχέσεις του με τα θέματα αυτά, δεν είναι πρωτόγνωρο για επενδυτές να αμφισβητούν μια νομοθετική ρύθμιση με διαφορετικούς τρόπους. Είναι δυνατόν να ξεκινήσει μια διαιτησία, αλλά παράλληλα με τη διαιτησία αυτή να υπάρξει αμφισβήτηση μιας νομικής ρύθμισης και σε εθνικό επίπεδο, δικαστικό επίπεδο, και αυτά είναι διαφορετικού τύπου θέματα και διαφορετικού τύπου προκλήσεις ε, που θα πρέπει να τεθούν σε σχέση με το ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αυτό δεν είναι κάτι που σε καμία περίπτωση θα αμφισβητήσει αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνουμε εμείς για την προστασία των επενδυτών στις χώρες τις οποίες δραστηριοποιούνται στα πλαίσια των διμερών συμφωνιών των διεθνών συγγνώμη συμφωνιών. Ε, ελπίζω να αναφέρθηκα στις ερωτήσεις σας σε όλες, αν τυχόν όχι θα επανέλθω. Ευχαριστώ, ελπίζω πως ναι. Τώρα ο εισηγητής, ο κύριος Ζαλεύσκη. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Και ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή για τις διευκρινήσεις που μας έδωσε. Νομίζω ότι ακολουθούμε την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή ότι υπάρχει ένα δεύτερο επίπεδο ενότητας και κατανόησης των προβλημάτων. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στα όσα είπε η Σκέλλερ, ότι πρέπει να βρούμε μία φόρμουλα ε, μέσω της οποίας μπορούμε να συζητήσουμε αυτά τα ουσιαστικά θέματα σχετικά με την προστασία των επενδύσεων που προσφέρουμε στους επενδυτές των τρίτων χωρών. Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση είναι χρήσιμη, διότι θα διευκρινίσει και, διευκρινίσει και τις προθέσεις της Επιτροπής για το μέλλον όσον αφορά τους επενδυτές. Αλλά δεν είναι το θέμα ακριβώς το οποίο συζητήσαμε. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να συζητηθεί σε αυτό το χρόνο. Θα διατυπώσω τις προτάσεις μου στην έκθεση, νομίζω την ερχόμενη εβδομάδα και προτού τις παρουσιάσω επισήμως, θα τις διανύμω μεταξύ των σχεδόν εισηγητών, ώστε να πούν τα σχόλιά τους και να μας βοηθήσουν και ώστε η συνεργασία να είναι όσο καλύτερα από την αρχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Αυτό το σχέδιο έκθεση θα συζητηθεί στην επόμενη Ολομέλεια το Φεβρουάριο. Moving to item 17. Ερχόμαστε τώρα στο 17. Επιτροπή θα είναι η υπεύθυνη, η αρμόδια Επιτροπή ε, για ε, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και γίνεται συζήτηση σε ανακοίνωση Επιτροπής σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ε, στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας. Ε, εδώ έχουμε να κάνουμε το σχέδιο έκθεσης, το έχετε μέσα στους φακέλους σας. Ο εισηγητής μας είναι ο Γιάννικ Ζαντό και τον παρακαλώ να παρουσιάσει την έκθεση, το σχέδιο έκθεσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρουσιάσετε το πλαίσιο αυτής της γνωμοδότησης που ήδη κυκλοφόρησε. Απλά και μόνο προς υπόμνησή σας, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμφισβήτητα εδώ και πολλά χρόνια είχε ηγετική θέση από πλευράς πολιτικής, ήταν αρκετά φιλόδοξη όσον αφορά τις ΑΠΕ και ε, για τις έρευνες και τη βιομηχανία. Η Ευρώπη έγινε ο ηγέτης ε, στο παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τις ΑΠΕ γνωρίζουμε ότι αυτή η κατάσταση εξελίσσεται, εξελίσσεται επειδή οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια έχουν γίνει ένα σημαντικό επενδυτικό κλάδο στα πλαίσια τη παγκόσμια οικονομία και ορισμένε χώρε άλλωστε έχουν αναπτύξει μεγάλες εμπορικές δραστηριότητες. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη από τα κράτη όσον αφορά τις ΑΠΕ για παράδειγμα στην Κίνα με τα φωτοβολταϊκά, αλλά επίσης μπορούμε να αναφέρουμε και την αιωλική ενέργεια και επίσης τη μεγάλη ανταπόκριση των Ηνωμένων Πολιτειών και αναμένεται από την Ευρώπη να κινηθεί σε αυτό το τομέα, να προχωρήσει σε έρευνες, να κάνει τη μελέτη της και να μας πει αν πράγματι υπάρχει dumping από πλευρά της Κίνας και ποιος μηχανισμός υπάρχει για να υπάρξει μια εμπορική άμυνα Λοιπόν, από τη δική μας άποψη, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να διατηρήσουμε αυτή τη φιλοδοξία όσον αφορά τους πολιτικούς στόχους, κλίμα ΑΠΕ, αλλά και όσον αφορά την βιομηχανική ικανότητα που έχει η Ευρώπη. Και αυτό σημαίνει πολλά πράγματα, ε, τα οποία βλέπουμε μέσα σε αυτή τη γνωμοδότηση. Επίσης, και αυτό έχει σχέση με τα όσα έλεγα για την περίπτωση της Κίνας, πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η Ευρώπη έχει πληκιστεί με τους απαραίτητους μηχανισμούς εμπορικής άμυνας, αν θέλετε, όταν υπάρχει αθέμετος ε, ανταγωνισμός. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο έχει σχέση με τις πρωτύτερες συζητήσεις που είχαμε για τις δημόσιες συμβάσεις και έχει σχέση με την τοπική διάσταση ε, του θέματος των ΑΠΕ. Γεγονό είναι ότι όταν βλέπει κανεί την οδηγία για τη ΑΠΕ, υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο, δηλαδή πώ μπορεί κανεί να ενισχύσει τι τοπικέ οικονομίε, πώ μπορούμε να ενισχύσουμε ε, την προμήθεια ΑΠΕ τοπικού επίπεδου με σκοπό να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, να υπάρξει μια πράσινη οικονομία που θα λαμβάνει υπόψη ε, και τη βιομηχανία και την κοινωνία. Ε, για παράδειγμα, αυτό σημαίνει, και το επαναλαμβάνω συνέχεια, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, σημαίνει δηλαδή ότι μέσα σε αυτά πλαίσια να χρησιμοποιήσουμε τις δημόσιες συμβάσεις για το σκοπό αυτό. Κάτι άλλο σημαντικό που συζητείται είναι το θέμα ε, των υδρογοναρθράκων, κατά πόσον αυτό μπορεί να ληφθεί υπόψη σημαντικά σε διεθνές επίπεδο. Και θέλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να ενσωματώσει αυτά τα στοιχεία. Όταν μετατρέπεται ένα πεδίο σε παραγωγής ε, υπάρχει εκείνο το οποίο λέμε έμεση αλλαγή ε, της χρήσης γης ε, στον υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για ορισμένε χώρε όπω η Ινδονησία, για παράδειγμα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, δεδομένου ότι οι εισαγωγέ πετρελαϊκών προϊόντων αντιπροσωπεύουν πάνω από 500 δισεκατομμύρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο ετησίως, πρέπει να αποφύγουμε όχι την ενίσχυση αυτής της ε, διάσταση των ΑΠΕ, αλλά να μειωθεί το εμπορικό μας ισοζύγιο, το εμπορικό μα ε, έλλειμμα, Και αυτό έχει σχέση με τι δημόσιε δαπάνε και τη δέσμευση της Ευρώπης μετά το G8 και το G20 να ε, περιορίσει τις επιδοτήσεις. Και ένα τελευταίο στοιχείο που θέλω να αναφέρω, που δεν ε, το μνημονεύω στις ε, περιορισμούς ε, που υπάρχουν εδώ, δηλαδή το θέμα των ΑΠΕ, των βιομηχανικών εταιρικών σχέσεων, συμπράξεων, σε συνεργασία με την περιοχή της Νότιας Μεσογείου. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσει για συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, μεγάλη της εμβέλειας και νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα μεγάλο κέρδος για την Ευρώπη και την Νότια Μεσόγειο, δηλαδή σε αυτές τις συμπράξεις να υπάρχει και ένα στοιχείο ισχυρό των ΑΠΕ. Ε, είμαι στη διαθεσή σας για να ακούσω τα σχόλιά σας, τις αντιδράσεις σας. Ευχαριστώ. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Ας ακούσουμε και τις άλλες ομάδες, αρχίζοντας από το ΕΛΚ, Κρίστοφερ Φιέρνα ή ο Ντάνιελ Κασπάρη. Ποιος από τους δύο θέλει. Κύριε Κασπάρη. Αγαπητοί συνάδελφοι, αντικαθιστώ τον σκιώδη εισηγητή και θα ήθελα να διαβάσω τα σχόλιά της. αρχίσω όμως με ένα προσωπικό σχόλιο. Όταν μιλάτε για τα προϊόντα, για τέτοια προϊόντα, θυμήθηκα τα προϊόντα από κοκοφίνικα που ήταν φιλικά ε, προς το περιβάλλον. Είναι εξαιρετικά ε, σημαντική, σημαντικός ο φάκελος αυτός. Σημερίζομαι τα περισσότερα από όσα υποστηρίζει ο εισηγητής και θα ήθελα να διευκρινίσω κάποια σημεία. Ενθάρρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσει μια δημιουργική προσέγγιση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι βέβαια σημαντικό οι μηχανισμοί να είναι προσαρμόσιμοι και εύπλαστη. Έπειτα είναι μεγάλη ε, σημασία τα SPI, αλλά πρέπει πάντα αυτά να γίνονται με στενή συνεργασία με τους άλλους αρμοδίους φορείς. Επίσης, συμφωνώ με αυτά που προτείνονται στην παράγραφο 3, ότι πρέπει δηλαδή να δοθεί έμφαση να παρέχονται κίνητρα για χρήση ανανεώσιμων πηγών και ιδίων πόρων. Επίσης, όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες, πιστεύω πως μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε, αλλά μόνο εκεί που είναι αναγκαίο. Παράγραφος 4, βιωσιμότητα. Να τονίσω ότι πρέπει να διασφαλίσουμε να είναι βιώσιμες και προσιτές, εφικτές οικονομικά. Οι Χρειάζεται να επιτευχθεί συμφωνία στο πρωτόκολλο του Κιώτο, το οποίο θα επηρεάσει κιόλα την κατασκευαστική βιομηχανία στην Ευρώπη. Επίση, είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι όταν καταρτίζεται νέα νομοθεσία που έχει σχέση με μείωση των εκπομπών, εμεί ω νομοθέτε πρέπει να λάβουμε υπόψη τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που αυτό μπορεί να έχει στη βιομηχανία μας και έτσι να αποφύγουμε την μετανάστευση των εταιριών μας στις τρίτες χώρες. <coughs> Ευχαριστώ πολύ. Ε, να πω ότι η Μαρία Κορέα είναι σκιώδης εισηγήτρια του ΕΛΚ. Συνάδελφε, ε, δεν θέλω να μιλήσω εκ μέρου τη ομάδα γιατί ίσω με περιορίσει αυτό, οπότε γι' αυτό άφησα τον κύριο Κασπάρη να μιλήσει. Καταρχά, να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τώρα να ασκήσω και κριτική. Αρχίζουμε λοιπόν από τα καλά και πάμε στα άσχημα. Διαβάζω το σημείο νούμερο 2 και έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι σκληρή και να χρησιμοποιήσει αυστηρά μέσα για να μας βοηθήσει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Νομίζω πως το μόνο που έχετε χάσει είναι ότι αυτός είναι ένας τομέα στον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη χρησιμοποιήσει τέτοια μέτρα μέσα. Συγγνώμη. Μέτρα για, για παράδειγμα ανεμογεννήτριες, ε, βιοντίζελ, εθανόλη από την Νότια Αμερική, ό,τι κάνουν αυτοί το κάνουμε κι εμείς. Αλλά νομίζω πως αυτό που θέλετε να πείτε είναι ότι πρέπει να το κάνουμε πιο διευρυμένα και στα φωτοβολταϊκά. Ας είμαστε όμως ειλικρινείς και ας παραδεχτούμε ότι εάν θέλουμε περισσότερο εμπόριο και αν θέλουμε να διευκολύνουμε το εμπόριο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν θα ήταν καλό να σκεφτούμε πώς θα στοχεύσουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με μεγάλη ακρίβεια. Μιλήσατε για επιδοτήσεις, αλλά Πόσες επιδοτήσεις νομίζετε πως πηγαίνουν στην εξόριξη πετρελαίου. Δεν έχουμε ρυθμιστικά και ελεκτικά μέτρα για να αποφεύγουμε το dumping. Στο πετρέλαιο, για παράδειγμα. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχουν ρυθμίσεις για το dumping και στα φωτοβολταϊκά. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς και ας παραδεχτούμε ότι έχουμε αρκετά μέσα καταπολέμησης ε, ανορθόδοξων πρακτικών. Μετά, σημείο 4 για, την, ε, για τα κριτήρια βιωσιμότητας και την αποψήλωση των δασών κτλ. Ε, με βρίσκουν σύμφωνο πολλά από αυτά τα σημεία, τα συμμερίζομαι, αλλά νομίζω εδώ ότι ποτέ δεν φτάνουν αυτά που ψηφίζουμε εδώ πέρα. Πέρυσι ή πρόπερσι ποτέ ήταν που ε, κάναμε νομοθεσία για παράνομη υλοτομία και του δεν θα πρέπει να εισάγουμε ξυλία που έχει υλοτομηθεί παράνομα. Και τώρα πάμε ακόμα παραπέρα. Πρέπει να βάλουμε δηλαδή την ε, υλοτομία μέσα στην εμπορική συμφωνία. Θυμάμαι μία συνάντηση με έναν εκπρόσωπο της Ινδονησίας, όπου συζητήθηκε συζητήθηκαν τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε με την χρήση της γης, της καλλιεργήσιμης γης. Αλλά το θέμα δεν είναι τόσο απλό. Διότι εκείνοι πιστεύουν ότι έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τον τρόπο που χρησιμοποιούν τη γη. Και εδώ οι πράσινοι έχουν κάπως υπεριαλιστικό ρόλο όταν τους λένε ότι όχι έτσι θα το χρησιμοποιήσετε τη γη. Είναι μια πρόκληση αυτό. Ας είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για κριτήρια βιωσιμότητας εν γέννη. Διότι μπορεί να το πιστεύουμε, να το νιώθουμε και ίσως πρέπει να δώσουμε προσοχή στα κριτήρια αυτά, αλλά μήπως θα έπρεπε να δώσουμε προσοχή σε αυτά τα πράγματα που είναι πραγματικά άσχημα και κακά, διότι τώρα διασπόμαστε λιγάκι και χάνουμε την ουσία κάνουμε δηλαδή κάποια πράγματα που βελτιώνουν αυτά που ήδη είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν κάνουμε τίποτα για, τα, για τους τομείς που έχουμε πραγματικά τεράστιο πρόβλημα. Και τέλος, πιστεύω πως πρέπει να προσθέσουμε κάτι που θέλω σημαντικό. Πάνω στην ε, συμφωνία για τις ε, τεχνολογίες πληροφοριών, η οποία πιστεύω ήταν θαυμάσια, όμως η εμπορική συμφωνία για το περιβάλλον πού είναι. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αυτή η γνωμοδότηση πρέπει να γίνει για το εμπόριο προς όφελος του περιβάλλοντος. Και μπορούμε να κάνουμε πολύ καλύτερα από αυτήν εδώ τη γνωμοδότηση, διότι δεν βλέπω πώς αυτό, με αυτό εδώ το κείμενο θα διευκολύνουμε την, ε, το εμπόριο στις ανανεώσιμες ε, πηγές. Έχω ακούσει πολλές φορές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λέει ότι είναι δύσκολο, όμως βλέπω τώρα ότι οι εταίροι μας έχουν ήδη γράψει έναν, καταρτήσει έναν κατάλογο και λένε με ορισμένα περιβαλλοντικά προϊόντα και αυτό είναι όλο και λένε όχι τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να διευκολύνουμε το εμπόριο και να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να επιστρέψουμε σε αυτό, να μην το ξεχάσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο πρόεδρος. Μπέρντ Λάνε. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Κάποιες παρατηρήσεις έχω να κάνω. Για Νίκ. Στην παγκόσμια αγορά, τα ευρωπαϊκά προϊόντα των ανανεώσιμων είναι γεγονός ότι είναι σε ηγετική θέση. Είμαστε πρώτοι. Έχουμε πολύ μεγάλο μερίδιο της παραγωγής από ανεμογεννήτριες, την εξάγουμε το 75% εξάγουμε. Έχουμε λοιπόν αυτόν τον ηγετικό ρόλο, ο οποίος βοηθά εμάς να προωθήσουμε την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και την κλιματική προστασία του περιβάλλοντος στον κόσμο και να προστατεύσουμε και τις θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Αυτός ο ρόλος πρέπει να ενισχυθεί ακόμα παραπάνω. Πρέπει να δώσουμε βάση εκεί. Να δούμε πώς θα ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τον ηγετικό μας ρόλο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολλά διαφορετικά συστήματα προώθησης. Από την άλλη όμως πρέπει να έχουμε και έναν στόχο, το στόχο δηλαδή του 20% ενέργειες από ανανεώσιμες. Και πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτά τα σύστηματα προώθησης, πόσο υπαρκούν, τι μπορούμε να κάνουμε μετά το 2020 διότι οι επενδύσεις μέχρι τότε πάει, θα έχουν εξατμιστεί. Δεν θα έχουν μείνει κονδύλια και πλησιάζει ο χρόνος. Γιατί μετά από τότε ο στόχος μας είναι το 45% ενέργειας από ανανεώσιμες και χρειάζεται να δώσουμε ένα καθαρό στίγμα και ένα σήμα στην παγκόσμια αγορά. Επιπλέον, Όσον αφορά την προώθηση της έρευνας, της επιστημονικής έρευνας, πιστεύω πως αυτό πρέπει να το δούμε. Διότι πέραν από τις ε, επιχορηγήσεις, όταν κάποιο προϊόν είναι μαζικής κατανάλωσης, έχουμε πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. πρέπει να δούμε τι κάνουμε σε αυτό, διότι έχουμε πολύ, μεγάλα, πολύ μεγάλο απόθεμα τεχνολογικής εμπειρογνωμοσύνης, αλλά τι γίνεται, έχουμε και επίσης πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Όταν θα έρθουν οι επενδυτές και οι ανταγωνιστές μας από την Κίνα, θα έχουμε πρόβλημα, δεν θα είναι πια τα πράγματα όπως είναι τώρα. Αυτά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι, ο κύριος Σόλτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω. Αλλά πιστεύω ότι αυτά που είπε ο κύριος Λάγκε δείχνουν ότι η προσέγγιση του κυρίου Ζαντό μας οφεί στο να σκεφτούμε πώς θα βελτιώσουμε τα πράγματα. Ο τίτλος της έκθεσης, η γνωμοδότηση, αναφέρεται στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Αλλά αυτό που πρέπει να δούμε είναι πώς εμείς θα ενισχύσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ενία αγορά. και έχουμε παραμελήσει την επιστημονική έρευνα. Είναι όντως, είναι γεγονός. Και πολύ σωστά αναφέρατε και τις ε, άλλες δυνάμεις, τις άλλες αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ανώσης, με άλλες ε, συνθήκες εργασίας, οι οποίες μπορούν να επωφεληθούν. Εμείς Όταν ασχολούμαστε με την ενιαία αγορά, δεν πρέπει να ξεχνάμε και την παγκόσμια διάσταση. Εάν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί στον τομέα των ανανεώσιμων και, των, και της παραγωγής τους, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ε, προϋποθέσεις και διαφορετικές ε, Διαφορετικέ προποθέσει ε, ε, για την εσωτερική αγορά, για την ενιαία αγορά και για εκτός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωση. Όχι. Πρέπει να τα συνδέσουμε αυτά και γι' αυτό για τα σημεία 1 και 2 που ανέφερες Γιάννη, θέλω να πω ότι έχουμε ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναπτύξουμε περαιτέρω την έρευνα και τη συνεργασία και τη σύνδεση και αυτό με, τι, με τις ε, αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ας μην σκεφτόμαστε μόνο το κέρδος, αλλά ας σκεφτούμε και πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε παγκόσμια. Τα προβλήματα που έχουμε στον οικονομικό τομέα είναι πάρα πολλά. Έχουμε την κρίση, έχουμε την ύφεση, όμως ταυτόχρονα έχουμε και το θέμα του περιβάλλοντος. Η έρευνα είναι κάτι που θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Και αυτό συνδέεται και με το δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεν είναι μακριά από αυτό. Δεν πρέπει να παραμεληθεί στη χάραξη πολιτικής μας. Γι' αυτό η γνωμοδότησή μας ίσως μπορούσε να το αναφέρει, να γίνει μια προσθήκη. Επίσης, να πω ότι πραγματικά πρέπει να σκεφτούμε και να δούμε πώς μπορούν να διοχετευτούν, να απολυθούν στην αγορά τα παράγωγα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. καθώς εξετάζουμε και όλες τις υπόλοιπες διαστάσεις, δεν πρέπει να ξεχάσουμε και αυτή. Και να σας πω ότι από πλευράς των πρασίνων θα επεξεργαστούμε αυτά που ανέφερα. Mr. House from... Ο κύριος Χάρης, από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση που ήταν πολύ χρήσιμο να ακούσουμε και τις προτάσεις που έγιναν και τη συζήτηση που ακολούθησε. Εμείς από πλευράς Επιτροπής θα θέλαμε να κάνουμε τρεις παρατηρήσεις σχετικά με το σημείο 2. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να αναφέρουμε ότι ο ρόλος μας είναι ενεργός στη διερεύνηση, αλλά υπάρχει αθέμητο εμπόριο κυρίως σε αυτό το τομέα Ήδη αναφέρθηκε ότι υπάρχουν ε, έρευνες ε, για ορισμένε τεχνολογίες και η Επιτροπή ξεκίνησε μία μελέτη. Ε, δηλαδή μπορείτε να χαιρετήσετε τη συνεχή δραστηριότητα της Επιτροπής που προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι το εμπόριο δεν θα είναι αθέμητο. Αλλά αυτή η δραστηριότητα της Επιτροπής είναι σε εξέλιξη. Το δεύτερο σημείο αφορά το 3, όπου χαιρετίζεται την τοπική διάσταση. Πράγματι υπάρχει μια τοπική διάσταση όσον αφορά την ανάπτυξη των ΑΠΕ και θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι λειτουργούμε ε, στον, ε, στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Και εδώ αναγνωρίζουμε ε, τα ωφέλη του διασυνοριακού εμπορίου. Όταν μιλάμε για τοπικά ωφέλη, πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι θέλουμε να αναπτύξουμε πόρου που να είναι αποτελεσματικοί από πλευρά κόστου στα πλαίσια τη ευρωπαϊκή αγορά. Τρίτο σημείο σχετικά με τον τριμερή διάλογο που παροτρύνεται την Επιτροπή να εισαγάγει στοιχεία κλιματικών αλλαγών. Και αυτό όμως πρέπει να πείτε πάλι ότι η Επιτροπή έχει κάνει την πρότασή σας και επαφείτε σε εσά να εξασφαλίσετε ότι αυτή η πρόταση θα γίνει δεκτή. Αυτά ήταν τα τρία σημεία που ήθελα να θίξω. Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και την Επιτροπή. Απλώς για να διευκρινίσω το θέμα του look, το θέμα δεν είναι σε μας να ορίσουμε πώς στην Ινδονησία χρησιμοποιούνται οι γέες. Απλώς και μόνο να, να βεβαιωθούμε ότι όταν υπολογίζουμε το ποσοστό του άνθρακα και το ποσοστό της αηφορίας, ας πούμε του κοφινικελαίου, ε, νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει η αλλαγή της χρήσης γης. Δεν μπορούμε να πούμε εμεί του Ινδονησίου πώ θα χρησιμοποιούν τη γη του, αλλά να είμαστε βέβαιοι ότι εμεί όταν αξιολογούμε ε, το οικολογικό στοιχεία ε, των βιολογικών καυσίμων, ότι όλα τα στοιχεία έχουν ληφθεί υπόψη. Γεγονό είναι όμω ότι το High Look είναι υποσυζήτηση στο Κοινοβούλιο. Επίση, με τα χαρά θα υπογράψω με τον συνάδελφο Φέλνερ μια τροπολογία για να ενισχύσουμε ε, τις επιχορηγήσεις για τα πετρελαϊκά προϊόντα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτά τα προϊόντα, αν δεν απατώμε, δεν ε, εισέρχονται ε, στους κανονισμούς του ΓΚΑΤ και του ΠΟΕ. Συνεπώ. δεν υπάρχουν διεθνείς κανόνες για το επίπεδο των δοκρατικών ενισχύσεων στον τομέα αυτό. Τώρα, carbon catch βεβαίω, αλλά πάλι το διακύβευμα είναι να αποφύγουμε το ball catch, δηλαδή να φροντίσουμε οι βιομηχανίε μα ε, που είναι ισχυρές, που έχουν μεγάλη ικανότητα καινοτομία και ανταγωνιστικότητα, ότι δεν θα μετεγκατασταθούν επειδή είναι θύματα του αθέμητου ανταγωνισμού. Και σε αυτό το θέμα και σε πολλά άλλο είμαι υπέρ της απελευθέρωσης των ανταλλαγών τεχνολογίας. Αλλά οι διαπραγματεύσεις στο ΠΟΕ ε, έχει σταματήσει εδώ και νομίζω ότι εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Επίσης θα υπογράψω μια τροπολογία αν θέλει ο Μπέρντ μαζί του ε, για το στόχο 45% ΑΠΕ μέχρι το 2030. Συμφωνώ απόλυτα. Τελευταία παρατήρηση αναφέρθηκε το φλεκτ. Κάθε φορά που υπάρχει μια συμφωνία φλεκτ είναι διμερής. Δηλαδή υπάρχει μόνιμη διαπραγμάτευση του φλεκτ με όλες τις χώρες που επιθυμούν να συμμετάσχουν. Εκεί ε, γίνονται λοιπόν συζητήσεις από αυτού είτε με αφρικανικές ε, χώρες της Λατινικής ε, Αμερικής ή της Ασίας. Με τα χαράς θα εξετάσω τα σχόλιά σας και σίγουρα η συζήτηση θα συνεχιστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για το διακύβευμα τη τοπική διάσταση. Άλλωστε δεν θα διαφεύγει ότι ορισμένα κράτη-μέλη είναι υπέρ τη τοπική διάσταση. Υπάρχει η γαλλική μόνιμη αντιπροσωπεία που είναι παρούσα και γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Υπουργό Ενέργεια θέσπισε ένα νόμο για τα φωτοβολταϊκά. Και υπάρχει μια ε, κοινοτική προτίμηση σε αυτή τη νομοθεσία, σε αυτόν τον νόμο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Προθεσμία λοιπόν. 28 του μηνός. Το μεσημέρι. Η υιοθέτηση θα γίνει στην τακτική μας συνεδρίαση του μηνός Φεβρουαρίου. Τελευταίο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το 18, Συμφωνία Ένωσης Κίνας, μια επιπλέον συμφωνία η οποία έχει σχέση με την είσοδο της Δημοκρατίας και της, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας γιατί βλέπουν τις, τους τρόπους ένταξής τους στην αγορά να αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα. Σόλτς. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να αναφερθώ στο συγκεκριμένο θέμα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη συμφωνία με τη Λαϊκή Κίνα. Πιστεύω ότι εμείς θα πρέπει να συνενέσουμε. Η λαϊκή δημοκρατία έχει το δικαίωμα να δει την αποκατάσταση των δικαιωμάτων της ε, μετά από την ε, ελαφρά χειροτέρευση μετά την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρωμανίας. Το 124 των ΓΚΑΤ προβλέπει ότι στόχος μιας ζώνης ελευθέρων συναλλαγών και μιας τελωνιακής ένωσης είναι η διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών και όχι ή η δημιουργια περαιτέρω εμποδίων. Στα πλαίσια λοιπόν των ε, διαδικασιών που προβλέπονται από τον ΠΟΕ πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτήν την συγκεκριμένη διεύθυνση Η διεύρυνση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνεισφέρει θετικά στις διαδικασίες του ΠΟΕ site. Και όταν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις ε, δύο περιπτώσεις, του να ανήκει δηλαδή κάποιος ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να βρίσκεται εκτός, τότε η διαφορά αυτή θα πρέπει να εξομαλυνθεί. Negotiations with the People's Republic of China resulted in the draft agreement in the form of η συμφωνία προωθείται στα πλαίσια της ανταλλαγής των επιστολών και τα προϊόντα τα οποία προβλέπονται σε αυτήν την αντισταθμιστική συμφωνία είναι μανιτάρια, σοκολάτες, είδη ζαχαροπλαστικής. Διαρωτώ με γιατί η Ευρωπαϊκή επέτρεψε, επέλεξε τα συγκεκριμένα αυτά άρθρα και προϊόντα, ειδικά τα μανιτάρια. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δικαίως ότι οι ποσοστώσεις οι δασμολογικές σαν αντισταθμιστικό μέσο είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος για την αποζημίωση κατά κάποιο τρόπο και την αποκατάσταση της μίας πλευράς η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας θα αλληλοενημερωθούν για την θέση σε ισχύ της συμφωνίας αυτής. και μετά από την τελευταία γνωστοποίηση θα τεθεί σε λειτουργία η συμφωνία αυτή και οι εταίροι θα ολοκληρώσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες λοιπόν χωρίς καθυστέρηση για να μην δημιουργηθούν στρεβλώσεις στις αγορές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν και τους σκιώδεις εισηγητές και ελπίζω το ταχύτερο δυνατόν να προχωρήσουμε σε, σε μια γρήγορη προσπάθεια να κλείσει το συγκεκριμένο θέμα από το ΕΛΚ, Βουίνκλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόκειται για μια κανονική τακτική διαδικασία συνένεσης, πρόκειται για μια αντισταθμιστική ρύθμιση τεχνικής φύσης στα πλαίσια των κανόνων του ΠΟΕ. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν έχει κανένα πρόβλημα και θα υποστηρίξει τη συγκεκριμένη πρόταση. Ζαντού. Εμπιστεύομαι τον εισηγητή, τίποτα άλλο η Επιτροπή. κ. Βερλέ, από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ίσως να προσφέρω κάποιες διευκρινήσεις. Τα πιο σημαντικά έχουν ήδη υποθεί από τον εισηγητή. Ίσως να υπενθυμίσω απλά πάρα πολύ σύντομα κάποιες γενικές παρατηρήσεις σχετικά με το 120. So, Σχετικά με το 24 λοιπόν γάμα άρθρο του ΓΚΑΤ. Στόχος του συγκεκριμένου άρθρου είναι η κατάληξη σε μια αμοιβαία και για τις δύο πλευρές ρύθμιση μετά από την αύξηση των δασμολογικών επιβαρύνσεων οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν αφορούν νέες ε, περιπτώσεις, αλλά αντισταθμίσεις για ζημίες λόγω επιπλέον δασμών που θα πρέπει να πληρώσουν για τις εξαγωγές ε, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται από τους κανόνες του ΓΚΑΤ. Μετά λοιπόν από τη διεύρυνση της Ένωσης το 2007, το συγκεκριμένο άρθρο, σύμφωνα με το άρθρο 24, έχει ισχύσει για την Κούβα, τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Αυστραλία, και έγινε μια αντίστοιχη συμφωνία επίσης για τις Ηνωμένε Πολιτείες και η τελευταία σε εκκρεμότητα συμφωνία αφορά την Κίνα. Το πακέτο αυτό το αντισταθμιστικό αφορά επίσης το σκόρδο και τα επεξεργασμένα μανιτάρια. Σε αυτά τα προϊόντα οι δασμοί είναι υψηλότεροι από ό,τι στην προηγούμενη περίοδο που είχαμε τότε διαπραγματευτεί με την Κίνα. Για το σκόρδο είναι ένας απλός μαθηματικός τύπος, βασίζεται στα διαφορετικά ύψη των τελών και στο ύψος των ποσοτήτων. ...2.370.000 τόνοι η ποσόστοση του σκόρδου για την Κίνα. Και υπάρχει μια αύξηση κατά 33.000 για τα μανιτάρια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσθέσει 800 τόνους στο ποσό των 28.850, δηλαδή ε, ένα 3% αύξηση. Για να διευκρινίσω ότι πέραν αυτής της αντιστάθμισης, η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης και την διαβεβαίωση του κεκτημένου του ΓΚΑΤ από πλευράς της Βουλγαρίας δηλαδή το δικό τους κεκτημένο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να το μεταφέρουμε στο ευρωπαϊκό αντίστοιχο. Και η συμφωνία αυτή είναι ένα νομικό μέσο για να γίνει αυτή η μεταφορά. Και στα πλαίσια της συμφωνίας αυτής λοιπόν αναφερόμαστε και σε 2.206 τόνους σοκολάτες, αντίστοιχες ποσότητες ειδών ζαχαροπλαστικής ή προϊόντων ζαχαροπλαστικής. Αυτές οι αντιστοιχμιστικές συμφωνίες αφορούν όλες τις χώρες και τις εισαγωγές σε όλες τις χώρες και οι αυξήσει της ποσοστώση αντιστοιχούν σε αυτές οι οποίες ίσχυαν πριν από την ένταξη των δύο αυτών χωρών. Δεν ξέρω αν υπάρχουν επιπλέον ερωτήσεις. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους εισηγητές για τα θετικά του σχόλια. Υπάρχει κάποιο τελικό σχόλιο? Όχι. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Προθεσμία. Είναι το μήνα Φεβρουάριο της τακτική μας συνεδρίαση και τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη συνάντηση είναι την 20 και 21 Φεβρουαρίου, 9 το πρωί. Ευχαριστώ.